Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Καλημέρα σας. Άρχονται οι εργασίες αυτής της συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Ω συνήθως, ε, στο πρώτο σημείο έχουμε την έγκριση της ημερησίας διάταξης ε, των εργασιών της Επιτροπής. Σήμερα στην ημερησία διάταξη Έχουμε σημεία που είναι πολύ σχετικά. Έχουμε τη συζήτηση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής και των τροπολογιών που παρουσιάστηκαν. Έχουμε τη συζήτηση για τις αναφορές κατά τη Συμφωνία Άκτα, την παρουσίαση εκ μέρου του διαμεσολαβητή του κ. Διαμαντούρο ε, για την τετήσια έκθεση του διαμεσολαβητή και επίσης έχουμε και την παρουσίαση της ε, Ειδικής Επιτροπής που ζητά το Κοινοβούλιο ο Ευρωπαίος Δημοσιολογητής. Ε, κατόπιν έχουμε και πάλι την ε, αναφορά για τα ευρωπαϊκά σχολεία, μια αναφορά σε σχέση με το λατομείο ασβεστόλιθου στη Γαλλία και μια της που αφορά τα βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια Αυστρίας και Γερμανίας. Ε, το πρώτο τμήμα της συνεδρίασης θα αφιερωθεί στην ψηφοφορία για τις δύο γνωμοδοτήσεις Όκεν και Γκέρικερ και κατόπιν θα έχουμε τη συζήτηση για την ετήσια έκθεση που έχει αναλάβει ο αδελφός Τσίτσεστερ και έχουμε και δύο γνωμοδοτήσεις ε, των κυρίων Βάλεαν και Σαλαβράκου και να σας υπενθυμίσω σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες ε, έχουμε και τη γνωμοδότηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα που θα ψηφιστεί στις 12 Ιουλίου. Προθεσμία για τις τροπολογίες έχει καθοριστεί στις 5 ε, Ιουλίου στις 5 το απόγευμα και σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση Σαλαβράκου ψηφοφορία 19 Σεπτεμβρίου τροπολογίες μέχρι τις 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα και σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση για την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχουμε την ψηφοφορία για τις 19 Σεπτεμβρίου και προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών 20 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα. Στην ε, ημερήσια διάταξη είδαμε ότι γύρω στις 10.30 θα ξεκινήσει η συζήτηση για τις αναφορές που έχουν να κάνουν με την Συμφωνία Άκτα και κατόπιν η Επιτροπή θα εξετάσει τις εκθέσεις για την επίσκεψη στο Βερολίνο και την έκθεση για την επίσκεψη στη Ρουμανία. Κατόπιν θα έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών στις 11.30 και από τις 3 και μετά ε, θα έχουμε τις ανακοινώσεις ε, σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών και κατόπιν θα ακούσουμε τον Ευρωπαϊκό Μεσολαβητή, τον κύριο Δημαντούρο. Θα είναι παρόντες και οι υπογράφοντες των αναφορών για τα ευρωπαϊκά σχολεία κατά τη Συμφωνία ΣΑΚΤΑ και σχετικά με το λατομείο στη Γαλλία. αν και οι αναφέροντες ε, που παρουσίασαν ε, την, ε, θα είναι μάλλον παρόντες και οι αναφέροντες σε σχέση με τις αναφορές που παρουσιάστηκαν για τον περικό μελητήριο Αυστρίας και Γερμανίας. Παρακαλώ, κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ για την ημερήσια διάταξη μια τροπολογία και μια επιθυμία. Η τροπολογία αφορά το 13, έκθεση για τις επισκέψεις στην Ρουμανία, εξέταση τροπολογιών και έγκριση. Θα ήθελα παρακαλώ να αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση, γιατί πρέπει να το συζητήσουμε ως ομάδα. Παρακαλώ να εγκρίνετε να αναβληθεί η συζήτηση του σημείου 13. Αυτό είναι το αίτημά μου και η παράκλησή μου ο συνάδελφο Μπουρλάνζ θα είναι μόνο το απόγευμα εδώ, οπότε θα παρακαλούσα να αναβάλουμε τη συζήτηση για την επίσκεψη στην, ε, στο Βερολίνο για το απόγευμα. Αν ε, δεν γίνεται θα έχουμε πρόβλημα γιατί ο συνάδελφο Μπουλάν ε, δεν μπορεί να είναι σήμερα το πρωί. Αλλά το ένα είναι αίτημα, το άλλο είναι παράκληση. Αν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εάν οι άλλοι συνάδελφοι μπορούν ε, να είναι παρόντες και θέλουν να συζητηθεί το πρωί. Το δεύτερο θέμα συμφωνώ. Σας ευχαριστώ. Η ημερήσια διάταξη περιέχει το σημείο 12. Όταν ε, συντάσσεται η ημερήσια διάταξη. Έχουμε αναλάβει όλοι δεσμεύσει. Εγώ δεν μπορώ να συμμετάσχω το απόγευμα, άρα επιμένω το, η ημερήσια διάταξη να μείνει ω έχει. Το σημείο 12 με ενδιαφέρει κυρίω. Ωραία, πολύ σύντομα τότε. Εντάξει, εφόσον είναι πρόβλημα, ε, δεν εμένω για το Βερολίνο, μπορεί να μείνει. Ε, μπορεί να μείνει το Βερολίνο, αλλά θα ήθελα να βληθεί η συζήτηση για την Ρουμανία. Μάλιστα θα το δεκτώ, αλλά κάποιες φορές έχουμε την εντύπωση ότι κάποια ομάδα εδώ θέτει όλους τους όρους ε, εργασίας σε αυτή την Επιτροπή. Και ε, να σας πω ότι το ΕΛΚ ε, <laughs> τώρα αν δεν μπορεί να σταθεί, θα πρέπει να ακολουθεί και όλη η Επιτροπή, τι να σας πω, είναι κάποιο διπραστικό. Όμω, ε, πραγματικά μου χρωστάτε πάρα πολλέ χάρε, Δεν είναι η πρώτη φορά. Bene, ε, allora. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ψηφίσουμε το πρώτο σημείο στην ημερησία διάταξη. Την έγκριση της ημερησίας διάταξης όπως τροποποιήθηκε. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Όχι. Εγκρίνουμε λοιπόν την ημερησία διάταξη και απλώς την επόμενη φορά θα συζητήσουμε την επίσκεψη στη Ρουμανία. Δεύτερο σημείο στην ημερησία διάταξη, ο συνήθως, έγκριση των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων. Πρέπει να εγκρίνουμε λοιπόν τα πρακτικά της 19 η Μαρτίου, 24 η Απριλίου και 8 η Μαου. Είστε υπέρ, υπάρχουν αντιρρήσει. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίνονται τα πρακτικά των τριών συνεδριάσεων αυτών που ανέφερα. Να σας ενημερώσω ότι ε, στο φύλλο της Προεδρίας επισυνάπτεται και προτάσεις να κλείσουν κάποιες αναφορές ε, ε, είτε γιατί δεν λάβαμε κάποια απάντηση από τους ε, αναφέροντες, ε, είτε γιατί κατέληξε η αξιολόγηση των αναφορών σε αυτό το συμπέρασμα. Από την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα επισυνάπτεται επίσης στο έγγραφα εργασίας και θα δίνεται εκ των προτέρων σε όλους τους συναδέλφους ένας κατάλογος που θα περιλαμβάνει τις αναφορές ή τις ε, αμφίβολες αν θέλετε αναφορές ή τα αμφίβολα ζητήματα που δεν ε, θεωρήθηκαν ότι εμπίπτουν στον κανονισμό ε, έτσι ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι να κρίνουν και οι ίδιοι τα θέματα αυτά και να ζητήσουν αν επιθυμούν να μπουν στο χρονοδιάγραμμα. Δεν έχω κάποια άλλη ανακοίνωση, έτσι λοιπόν αν δεν ε, ζητεί κανεί το λόγο θα περάσουμε στο σημείο 5 να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Έχουμε την ψηφοφορία για την πρώτη γνωμοδότηση. Στο σημείο 5 έχουμε τη γνωμοδότηση για ε, το νόμο περί δικαιωτικής δικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Όκεν, παρακαλώ, έχει το λόγο για την παρουσίαση. Θα μιλήσω δανέζικα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα με παρακολουθήσετε, θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την συμβολή τους σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Ελπίζω επίσης να επιδείξετε κατανόηση στο γεγονός ότι ήταν δύσκολο να περιλάβουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση όλα τα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να το συζητήσουμε επανειλημμένα. Εάν περάσει αυτό το θέμα, επίσης και από την Νομική Επιτροπή, θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος για τους Ευρωπαίους πολίτες διότι η αρχή ότι η δημόσια διοίκηση πρέπει να παρέχει υπηρεσίες που είναι γνωστή σε πολλές χώρες όπου η διοίκηση είναι στην υπηρεσία των πολιτών και δεν ασχολείται κυρίως με την διοικητική πλευρά της δουλειά της, την εσωτερική, είναι πολύ σημαντική. Γιατί πολύ συχνά ε, το να μην ασχολείται κανείς αρκετά με τους πολίτες ε, είναι για να προστατεύσει η διοίκηση των εαυτό της. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ο πολίτης να, ξαναπεί, να ξαναμπεί στο κέντρο. Η πείρα που έχουμε από αυτό είναι πολύ καλή και πιστεύω ότι με αυτή την πείρα οι διοικήσεις μπορούν να βοηθήσουν όλους τους πολίτες βέβαια να εφαρμοστεί η κουλτούρα αυτή η διοικητική σε όλες τις χώρες θα ήταν ένα μεγάλο βήμα. Πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη κατάσταση πνεύματος. Είναι μια πολιτιστική αλλαγή πραγματικά. Ελπίζω λοιπόν να εγκριθεί αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης Ελπίζω να μπορέσει να επιδράσει και στα πλαίσια της σύνταξης του νέου κανονισμού. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μία διαμάχη επί του θέματος αυτού με το Συμβούλιο διότι δεν είναι προφανές ε, πώς θα υπάρξει αυτή η αλλαγή. Δεν έχει περάσει ακόμη και στην, ε, στην νομοθεσία της Ένωσης. Ελπίζω όμως να αποτελέσει ένα μεγάλο βήμα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κυρία Όκεν για τις εργασίες που αναλάβατε και ελπίζουμε και εμείς να βγουν ελευθερινά τα όσα ευχηθήκατε στην πρέμβασή σας. Να ξεκινήσουμε τη ψηφοφορία για την έκθεση Όκεν. Να περάσουμε λοιπόν στη ψηφοφορία της ε, πρώτης ε, παραγράφου, 2, πρώτη προλογία, παράγραφος 2, Μπασέσκου. Ε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 3, Έλληνα Μπασέσκου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3, Μπέκερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 4, συγγνώμη, τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 5, Μπασέσκου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 6, Μπέκερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 8, Μπασέσκου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Καταπίπτει. Γιατί εγκρίθηκε η προηγούμενη τροπολογία, μόλις ψηφίσαμε. Περνάμε στην τροπολογία 9 Μπασέσκου, υπέρ, κατά. Εποχές. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, γιατί δεν σηκώσετε το χέρια σας. Τροπολογία 9 Μπασέσκου, για την παράγραφο 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10, όκεν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, παράγραφος 8, Μπέκερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, παράγραφος 9, Μπέκερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13, παράγραφος 10, Μπέκερ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10, τροπολογία 14, όκεν, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15, παράγραφος 11, βαλέσα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16, παράγραφος 12, βαλέσα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17, παράγραφος 12, μπέκερ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18, παράγραφος 12, Μπασέσκου, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19, παράγραφος 12α, νέα. μπέκερ, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20, στην παράγραφο 12β, νέο. μπέκερ. Εδώ ζητείται η τμήματική ψηφοφορία. Να ψηφίσουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Δεν πρέπει να ελέγξουμε. Μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Για το πρώτο τμήμα έρχεται ψηφοφορία υπέρ. κατά απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται τροπολογία 21 Μπέκερ υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται Ψηφίζουμε την γνωμοδότηση στο σύνολό τη. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Ευχαριστούμε την κυρία Όκεν. Να περάσουμε στο δεύτερο σημείο, γνωμοδότηση σχετικά με την 28η έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Η κυρία Γκέριγκερ είναι η συγγήτρια. Παρακαλώ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές γιατί ήταν εξαιρετική η συνεργασία μας. Ήταν πάρα πολύ καλές και οι προτάσεις τροπολογιών. Οι περισσότερες από αυτές προτείνω να τις δεχθούμε. Είχα κάποιες αμφιβολίες, μερικές τροπολογίες ε, που αποδυναμώνουν το κείμενο θεωρώ ότι πρέπει να καταψηφιστούν, αποδυναμώνουν τις ε, γενικές ε, προτάσεις που κάνουμε σε σχέση με τη βελτίωση της ε, εφαρμογής νομοθεσίας στο μέλλον. Οπότε παρακαλώ πολύ, λίγη προσοχή. Ελπίζω ότι τις απόψεις μου θα τις δεχθεί και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Ήμουν εισηγήτρια και στην Επιτροπή Νομικών ε, Θεμάτων για το θέμα αυτό και ήταν ε, περίπου ίδια η προσέγγιση ε, και η ίδια προσέγγιση προτείνω και τώρα. Ευχαριστώ πολύ και ας περάσουμε στην ψηφοφορία, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ευχαριστούμε την κυρία Γκέριγκερ, ελπίζουμε να μην υπάρχουν προβλήματα. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν και για την γνωμοδότηση αυτή. Λοιπόν, τροπολογία 1, Μπασέσκου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, παράγραφο 5, Βέρτμαν, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, παράγραφος 7, Μπασέσκου, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, παράγραφος 7α, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. για να ελέγξουμε. Να ξαναψηφίσουμε για την τροπολογία 4. Ε, Κυρία Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, Έχουμε κάποιε αμφιβολίε σε σχέση με τις τροπολογίες 3 ε, με τη σχετική ψηφοφορία. Μπορούμε να επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία για την τροπολογία 3 γιατί δεν είμαι σίγουρη ε, ότι ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ για το έτοιμά σας, ε, γιατί ναι, μου είπαν ότι δεν ήταν σαφής η ψηφοφορία. Εγώ νομίζω ότι εγκρίθηκε. Αν συμφωνούν τώρα λοιπόν και οι συνάδελφοι, να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, χωρίς μικρόφωνο η Πρόεδρος. Ξαναψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 3, Μπασέσκου, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 στην παράγραφο 7α. Οκ. Okay. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Στην παράγραφο 8. Μπέκερ. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 στην παράγραφο 8 Μπασέσκου. Υπέρ. Κατά. εποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 στην παράγραφο αλφα Μπέκερ. Υπέρ. Κατά. εποχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 στην παράγραφο 9 Μπασέσκου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είμαι σίγουρη. Να επαναλάβουμε την ψηφορία για τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Εννέα, ναι, ε, εννέα. Εννιά, εννιά. Εννιά υπέρ, εννιά κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Απορρίπτεται η τροπολογία αυτή. Τι σημαίνει να number Nine to nine, yes. It was. So it falls. That's right. The amendment. No, it was this one. No, we're on this one. That was nine. Now we're on paragraph 11, amendment nine by Mrs. Alkin. So. Allora, viene respinto. Απορρίπτεται λοιπόν. Κατόπιν διαβούλευση και με την γραμματεία και να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Τροπολογία 9 στην παράγραφο 11. Όκεν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 στην παράγραφο 12. Όκεν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 στην παράγραφο 12α. Όκεν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12, όκεν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ξαναψηφίσουμε. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να το δούμε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Όχι. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. Τροπολογία 13 για την παράγραφο 13. Όκεν υπέρ. Κατά. εποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 για την παράγραφο 14α. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση στο σύνολό τη. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στη συνάδελφο. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε τις ψηφοφορίες. Και να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Έχουμε την ετήσια έκθεση που έχει αναλάβει ο συνάδελφος Τσίτσιστερ, αλλά δεν βλέπω να παρευρίσκεται. Να ζητήσω από τη συνάδελφο Βάλεαν να μήπως ε, θα μπορούσαμε να δούμε το δικό της σημείο. Μάλιστα, έτσι λοιπόν θα σας δώσω το λόγο στο σημείο αυτό για την γνωμοδότηση σχετικά με το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και την ηθαγένεια για την περίοδο 2014-2020. Ευχαριστώ κύριε Βάλεαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εξετάζουμε τις τροπολογίες της, τους πρότασης κανονισμού για ε, τα δικαιώματα της ηθαγένειας 2014-2020. 48 τροπολογίες ε, κατατέθηκαν. Τα βασικά ζητήματα των τροπολογιών ε, είναι τα εξής. Πρώτο, Διακόπτει η Πρόεδρος. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τη διερμηνία. Εντάξει, μπορώ να συνεχίσω. Ακούτε? Ωραία. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ένα από τα πρώτα θέματα που θέτουν οι τροπολογίες είναι η ενίσχυση για τα ζητήματα ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης της βίας και την εφαρμογή ε, της ε, σύμβασης ε, των ατόμων με αναπηρίες. Πρέπει οι στόχοι να διατυπωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να υπερβαίνουν την καταπολέμηση των διακρίσεων και να συμπεριλάβουν την προώθηση της ισότητας και των δημοσιο... δικαιωμάτων, ειδικότερα για το θέμα της ομοφιλοφιλοφοβίας ε, και του ρατσισμού που πρέπει να είναι ένα τμήμα του προγράμματος. Τα θέματα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να θεωρείται μια ανεξάρτητη πολιτική του προγράμματος και η καταπολέμηση της βίας πρέπει να αναφέρεται ως στόχος, όπως επίσης και η ε, πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των μικρών παιδιών. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι στόχοι που προσπαθούμε να τους επιτύχουμε Έχουμε με διάφορους τρόπους μέσω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η προώθηση της ισότητας των φύλων και η καταπολέμηση της βίας θα είναι υποφελής ε, για όλους όσους είναι θύματα διαφόρων ειδών ε, ε, ρατσισμού και βίας. Ε, επίσης, ε, η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχει, γιατί είναι ένας σημαντικός τομέας, παρέχει υπηρεσίες που συμπληρώνουν τις κυβερνητικές υπηρεσίες και ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα και ανησυχίες που εκφράζονται ε, από όσους ε, εκπροσωπούνται με αυτόν τον τρόπο σε όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις. Θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε την ποιότητα της νομοθεσίας θέλοντας να δώσουμε περισσότερα στοιχεία και δεδομένα τα οποία με διαφορετικό τρόπο δεν θα φτάσουν στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Θέλουμε επίσης να αυξήσουμε τη δημοκρατική νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εφαρμογή ε, της νομοθεσίας ε, και σε ό,τι αφορά την επίλυση διαφορών σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ε, στο άρθρο 5 παράγραφος 2 ζητώ την υποστήριξη των μη κυβερνητικών οργανισμών που διεκπεραιώνουν δραστηριότητες του προγράμματος. Επίσης, υποστήριξη ε, ορισμένων ε, ευρωπαϊκών και εθνικών δικτύων, των οποίων οι δραστηριότητες έχουν να κάνουν με τους στόχους του προγράμματος. Και τρίτο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι τροπολογίες ε, είναι η διαφορετική ειδικοί στόχοι του προγράμματος ε, κατά πόσο θα πρικοδοτηθούν με τα απαραίτητα κονδύλια ετησίως. Δεν αναφέρονται στοιχεία σε σχέση με την κατανομή των κονδυλίων στις διάφορες δράσεις και προτεραιότητες ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι τα επίπεδα των κονδυλίων θα προβλέπονται κάθε χρόνο η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, κατά πολέμηση βίας ε, κατά των ε, γυναικών, των παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων ε, επιζητούν κονδύλια κάθε χρόνο και τα δίκτυα που εργάζονται επί των ζητημάτων αυτών πρέπει να έχουν επαρκή χρηματοδότηση για να μπορούν να συνεχίσουν την δουλειά τους με αποτελεσματικό τρόπο. Το νομικό κείμενο του προγράμματος πρέπει να περιλαμβάνει περιλαμβάνει κάποια στοιχεία που να δείχνουν ότι κάτι τέτοιο θα συμβαίνει κάθε χρόνο, ότι θα υπάρχουν ε, τα κονδύλια αυτά. Κάποια ε, πράγματα θα ήθελα να πω για τις τροπολογίες. Ε, η έγκριση της γνωμοδότησης προβλέπεται τον Ιούλιο, 12 Ιουλίου συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Βάλεαν. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της, στην εκπρόσωπο της Επιτροπής, την κυρία Σρίτερ. Thank you, Mr. President. Um, Ευχαριστώ πολύ. Πολλές από τις τροπολογίες που προτείνονται συμπορεύονται απολύτως με, την, με τις δικές μας προθέσεις, ισότητα φύλων, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, των παιδιών, των νέων, υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Όλα αυτά είναι ζητήματα ε, τα οποία καλύπτονταν από την αρχική μας πρόταση, ενδεχομένως όχι ε, με ε, επαρκώς σαφή τρόπο, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ε, ιδιαίτερες αντιρρήσεις. Ε, για ποιο λόγο να μην είναι πιο ε, σαφή και πιο ορατά τα θέματα αυτά στην πρόταση, δεδομένου ότι είχαν ήδη συμπεριληφθεί στο αρχικό μας κείμενο. Οπότε ουσιαστικά επικροτούμε περαιτέρω διευκρινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Βαλέσα τώρα. Έχετε το λόγο κύριε Βαλέσα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τη συντάκτρια της γνωμοδότησης. Είναι αντικειμενική η γνωμοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό διότι προωθεί θέματα που αφορούν την ε, ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Και βεβαίως αναφέρεστε και είναι πολύ καλοδεχόμενο, καλοδεχούμενο αυτό και στην οικονομική πλευρά είναι πολύ σημαντικό για προγράμματα που αναλαμβάνουν μικρές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Δεν είναι επίμαχες οι περισσότερες τροπολογίες, αλλά δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε όλες, υπέβαλα εγώ ίδιος πέντε τροπολογίες και κυρίως ε, μιλάω για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού, καλύτερη συνεργασία σε περιφερειακό, τοπικό και εθνικό επίπεδο και Πρέπει επίση να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα με ειδικέ ανάγκε μπορούν να απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων του ω πολίτε τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κάσμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπω πάντα, με χαρά συνεργάζομαι με την κυρία Βάλιαν για οποιαδήποτε θέματα που απασχολούν την Επιτροπή μας. Χαίρομαι για την στεναρή και συνολική στάση που ανέλαβε, διότι θα υπάρξει μια ενοποίηση τριών ήδη ε, λειτουργούντων προγραμμάτων. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει σαφήνεια και να εμείνουμε στη γνωμοδότηση ότι το πρόγραμμα πρέπει να καταρτιστεί με πολύ προσοχή, όπως είπε και ο κύριος Βαλέσα και η κυρία Βάλιν, γιατί αφορά και έχει επίδραση στους ε, πολίτες μας. Ε, Βεβαίω θα συνδυάσουμε τρία προγράμματα δικαιωμάτων και ηθαγένεια. Θα απλοποιήσουμε τα πράγματα και περισσότερη συνέπεια στην πολιτική μας. Αλλά κάθε πρόγραμμα πρέπει να διατηρήσει τους ειδικού του στόχους για να υπάρξει συνολική και αποτελεσματική προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών που πηγάζουν ακριβώς από την ε, ηθαγένεια της Ένωσης. Υπέβαλα τροπολογίες. Μήπως θα ήταν δυνατόν Κοιτάξτε, ήμουνα ηθοποιός και αν κάποιος ψιθύριζε στην τελευταία σειρά του θεάτρου θεωρούσε ότι θα έλεγαν τι χάλι ηθοποιός είναι, οπότε με ενοχλούν οι ψήθυροι. Μα δεν λέγαμε αυτό, λένε οι συνάδελφοι του κ. Κάσμαν. Λοιπόν, επανέρχομαι στη γνωμοδότηση, πολύ πιο σημαντικό. Νομίζω ότι επιτυχάνουν την αναγκαία ισορροπία μεταξύ διαφορετικών απόψεων οι τροπολογίε. Μιλάμε για την καταπολέμηση των εγκλημάτων τη αλλοδοξία και τη βία και ιδιαίτερα σε σχέση με το πρόγραμμα Δάφνη. Θαυμάσια λοιπόν η εργασία της ηγήτριας. Επαναλαμβάνω αυτό που είπε και η κυρία Βάλεαν. Ζωτική σημασία είναι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να έχουν βεβαιότητα για την εφαρμογή και συνεχιζόμενη χρηματοδότηση για να μπορέσουν να προγραμματίσουν την εργασία τους. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να υπάρξει μια αντικειμενική και δίκαια ε, παροχή χρηματοδοτήσεων στις μη κυβερνητικέ οργανώσει για να υπάρχει μια συνέχεια στη δουλειά τους, να υπάρχει μια σιγουριά ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Και οι τροπολογίε και η γνωμοδότηση βοηθάνε το πρόγραμμα, προσθέτουν νέους στόχους και την καλωσορίζω. Γιατί νομίζω ότι αποστέλει στους πολίτες μας το σωστό μήνυμα. Δύο σχόλια. Επειδή μιλάμε για τα γενικά δικαιώματα της ηθαγένειας, αναφέρουμε τη συνθήκη για, των Ηνωμένων για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικέ ανάγκε. Πολύ σημαντικό αυτό. Και προσθέτω για ενημέρωση στην Επιτροπή μα. Ανησύχησα πολύ την προηγούμενη εβδομάδα όταν έμαθα ότι το Κοινοβούλιο δεν κάνει αρκετά για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Χαίρομαι λοιπόν που μιλάμε για τη Σύμβαση των Ηνωμένων αν χρειάζεται να αναφέρουμε μόνο μία σύμβαση. Θα ήθελα αν είναι δυνατόν κάποιου είδους ορισμό τι εννοούμε όταν μιλάμε για το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γιατί ο καθένας ε, το ερμηνεύει όπως θέλει, κατά το δοκούν. Και η τροπολογία 5, εφόσον μιλάει για την αποδοχή διαφορετικών απόψεων, αλληλεγγύη και ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν θα πρέπει να μιλάμε καλύτερα για ισότητα για όλους είναι περισσότερο ερωτήσεις γιατί νομίζω ότι είναι θαυμάσια, αντικειμενική και στεναρή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Κάσμαν. Δεν ξέρω αν η κυρία Βάλεαν θέλει να ξαναπάρει το λόγο. Όχι. Εξαντλήσαμε λοιπόν αυτό το σημείο σήμερα. Να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 12 Ιουλίου, στη συνεδρία στις 12 Ιουλίου λοιπόν. Και καθώς ήρθε και ο συνάδελφος Τσίτσεστερ, να επανέλθουμε στο σημείο 7, θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσίτσεστερ για την ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που καθυστέρησα αλλά προσπαθούσα να κάνω το αδύνατο να επιτελέσω όλα τα καθήκοντα. Ε, βέβαια ξέρω ότι οι γυναίκες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό αποκλειστικά να τα καταφέρουν σε πολλά. Έχουμε 110 τροπολογίες για την έκθεση αυτή. Είχαμε μία προκαταρκτική συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία. Εργαζόμαστε επί μια σειρά συμβιβαστικών τροπολογιών. Έχω κάποιες ε, ήδη σε σχέση με την αφορά στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το πώς ε, θα αναπτύξουμε τις δημοκρατικές αρχές, ε, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία για το θέμα των μη παραδεκτών ε, αναφορών. Επίσης, πρέπει να θυμίζουμε στον εαυτό μας ότι μεγάλο αριθμό αιτήσεων επικεντρώνονται στο περιβάλλον, στη δικαιοσύνη και στην εσωτερική αγορά, στα συστήματα αυτά λοιπόν. Και πώς θα προωθήσουμε το ρόλο και τις ευθύνες της Επιτροπής μας, κυρίως σε ό,τι αφορά την ικανότητά της να ακούσει μάρτυρες και να υλοποιεί έρευνες. Εργαζόμαστε λοιπόν επί των θεμάτων αυτών. Είναι νομίζω ορθό να πω ότι η πλειονότητα των τροπολογιών θα είναι αποδεκτές. Έτσι λοιπόν θα διευρυνθεί κατά κάποιο τρόπο η έκθεση. Και έχουμε και σήμερα το απόγευμα μια ακόμη συνεδρίαση με τους κοιόδης εισηγητές. Πέραν αυτού δεν ε, είμαι έτοιμος να μπω τώρα σε λεπτομερή σχόλια για κάθε τροπολογία. Νομίζω ότι θα προέτρεχα. Το καλό θα ήταν να ακούσω τους συναδέλφους ε, αν έχουν κάποιες συγκεκριμένες ε, ανησυχίες ή αν θέλουν να υποβάλουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστούμε κύριε Τσίτσεστερ. Λοιπόν, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Uh, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να δω κύριο Βίλαντ, γιατί ήθελα να το ρωτήσω για την τροπολογία 65 για θέματα νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αλλά θα ψάξουμε αλλιώ να το μάθουμε. Είναι η δική σας επιτροπή ε, για τις δικές δραστηριότητες. Δεν χρειάζεται πολλά να ακούσετε από μένα. Κοιτάζοντας τροπολογίες, ε, συμφωνώ με αυτό που είπε ήδη ο κύριος Τσίτσεστερ είναι προφανές ότι οι περισσότερες θα τύχουν ευρεία ε, σε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Φλόιντ. Ο κύριος Κάσμαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλώς ορίζω την έκθεση του κυρίου Τσίτσεστερ. Εξαιρετική έκθεση και όπως είπα νωρίτερα νομίζω ότι καλύπτει ορισμένα θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Παραδείγματο χάρη την ελευθερία, την ελευθερία κυκλοφορία, τους Ρωμά και άλλες μειονότητες, τις διακρίσεις και την ισότητα των φίλων και επίσης ε, θέλω να αναφέρω ειδικά το θέμα των ατόμων με ειδικέ ανάγκες, ε, καθώς δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να χαιρούν ε, των ίδιων δικαιωμάτων. Όπως είπε και η κυρία Βάλεν προηγουμένως και νομίζω ότι όσα κάνουμε συμφωνούν με όσα έχουμε συμφωνήσει σε άλλες εκθέσεις. Όσο περισσότερη συνέχεια έχουμε για τα δικαιώματα των πολιτών τόσο το καλύτερο. Έχω προσθέσει μια τροπολογία που τονίζει τα εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία για ε, τα ζευγάρια του ίδιου φίλου και επίσης ε, αναφερόμαστε και στα θεμελιώδη δικαιώματα των LGBT στην Ευρώπη των ΛΟΑΔ στην Ευρώπη. Επίσης, ε, ε, θέλουμε να υπάρχουν διακρίσεις ε, απέναντι στου Ρωμά και σε άλλες εθνοτικές ομάδες, αλλά και σε ανθρώπου λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που υποστηρίζουν την προσέγγιση αυτή σε σχέση με ένα επίμαχο ζήτημα, δηλαδή το δίκαιο ιδιοκτησία ε, στην Ισπανία και συγκεκριμένα για το Λέιδε Κώστε για την ομολογία, ε, την ομοθεσία συγγνώμη, για την παράκτεια ζώνη. Όπω ε, ξέρετε, έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα από την Ισπανική κυβέρνηση και ελπίζουμε ότι θα υπάρχει μια δίκαιη επίλυση για του χιλιάδε ανθρώπου που απευθύνθηκαν σε εμά και πλήττονται από αυτή την ομοθεσία για την παράκτεια ζώνη όμως ε, καλωσορίζω την ε, κάθετη στάση που παίρνει ο κύριος Τσίτσεστερ στην έκθεσή του. Αν θέλουμε να μας πάρουν σοβαρά, θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ισχυρή θέση. Βλέπουμε ε, τα τελευταία έτη κάποιες ομάδες ε, μπορεί να παρουσιάζουν κάποια επιχειρήματα ίσως ε, για να περιορίσουν ε, την ισχύ της δικής μας άποψης στο Κοινοβούλιο, εγώ δεν θα συμφωνούσα με κάτι τέτοιο. Αν ε, δεν επιμένουμε και αν δεν είμαστε συνεπείς στην εφαρμογή της αρχής, τότε υποσκάπτουμε την ίδια την αρχή. Έτσι λοιπόν, πολύ καλή δουλειά. Είμαι σίγουρος βέβαια ότι θα υπάρχουν ε, και κάποιες αντιρρήσεις και άλλες τροπολογίες, αλλά εγώ καλωσορίζω το έργο σας και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας. Και όπως είπα και στην αρχή, η εκθέση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστώ, Μέγερ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσίτσεστερ για την έκθεση αυτή. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία επαναλαμβάνει το πόσο σημαντική είναι αυτή η Επιτροπή για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και για τους πολίτες γιατί αποτελεί φερέφωνο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί εκπρόσωπο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο της κρίσης που βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα θα έχουμε πολύ περισσότερες αναφορές και έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να μπορούμε να απαντήσουμε όπως πρέπει στα ζητήματα που θα μας θέσουν. Και εγώ παρουσίασα κάποιες τροπολογίες σε σχέση με το πόσο σημαντικό ε, εκεί είναι η συνεργασία ε, αυτής της Επιτροπής με τον ε, ίδιο ε, το Κοινοβούλιο με τις αρχές των κρατών μελών όπως και με το διαμεσολαβητή και επίσης ε, υποστηρίζω ότι μπορούν να υπάρχουν και άλλα συμπληρωματικά εργαλεία που έχουν ε, στη διάθεσή τους οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν δηλαδή να παρουσιάσουν κάποιες καταγγελίες στον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα θα τεθεί σε ισχύ σε λίγο καιρό η, η νομοθεσία για την πρωτοβουλία των πολιτών και αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα έχουν ένα άμεσο εργαλείο για να μπορούν να, να παρουσιάσουν θέματα που είναι σημαντικά για αυτούς και η Επιτροπή αυτή θα ήθελε να είναι χρήσιμο αυτό το μέσο. Σε ό,τι αφορά τώρα την ομοθεσία για την παράκτια ζώνη, έχω μια τροπολογία όπου αναφέρομαι ότι πρέπει να προστατεύσουμε την παράκτια ζώνη αποτελεσματικά και επίσης αναφέρομαι και ε, στις αντιφάσεις ε, που επέφερε η νομοθεσία τη ε, της ζώνη ζώνης και όπως είδαμε στη συζήτηση που είχαμε με την Ισπανική κυβέρνηση αυτή η θα πρέπει να επιλύσει δύο θέματα. Την προστασία της παράκτιας ζώνης, το δημόσιο χαρακτήρα της αφενός και αφετέρου να εγγυηθεί ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας για την παράκτεια ζώνη να ε, μην γίνει με αυθαίρετο τρόπο. Σας ευχαριστώ κύριε Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ κύριε Μέγερ. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσίτσεστερ για την έκθεσή του, που είναι εξαιρετική. Πολλές προτάσεις τροπολογιών υπήρξαν και εναγωνίως περιμένω τις ε, συνεδριάσεις, τις οποίες θα μπορέσουμε να τις συζητήσουμε. Οι δικές μας τώρα προτάσεις των πρασίνων. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να είναι μια πραγματική προστασία το Natura 2000 και στις διάφορες ε, αναφορές, διάφορες καταγγελίες ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει απώλεια βιοποικιλότητας ε, στις περιοχές αυτές, οι οποίες είναι περιοχές στις οποίες πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι τα πτηνά, η πανίδα προστατεύεται και από τους υπόλοιπους και από εμά αν οι υπόλοιποι δεν μπορούν να το καταφέρουν. Θα ήθελα επίσης ε, να σας επιστήσω την προσοχή στο εξής. Στην ε, δανική εκδοχή των τροπολογιών ε, υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει λέει το ακριβώς αντίθετο με την αγγλική εκδοχή. Φαντάζομαι ότι το σημειώσατε. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι θα έπρεπε να γίνονται και επιτόπου έλεγχοι. Θα ήταν εποφελές αυτό. Να πηγαίνουμε δηλαδή στις περιοχές αυτές και όχι ε, από μακριά να προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Οι ηλεκτρονικές ε, καταγγελίες είναι κάτι σύγχρονο, δουλεύει καλά και είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να ε, το λάβουμε υπόψη, ενδεχομένως να το προβλέψουμε. Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις τροπολογίες, γιατί ούτω ή άλλως θα τις ε, ε, συζητήσουμε και στις άλλες μας συνεδρία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάντως και να δούμε τι θα γίνει και με την νομοθεσία για την παράκτεια ζώνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Γιάρ. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Τον εισηγητή, συγγνώμη. Νομίζω ότι η δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών δεν θα πρέπει να δημιουργεί μεγάλες ε, διαμάχες μεταξύ μας. Βεβαίως ε, είναι το επισκεπτήριό μας αυτή η έκθεση. Αναφέρουμε στους άλλους ε, τι κάνουμε. Βεβαίως ο καθένας μας από ομαδες ομάδα δίνει άλλο βάρος σε κάθε θέμα αλλά πρέπει οπωσδήποτε να καταλήγουμε σε κοινούς παρονομαστές και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι στόχος μας να εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία η έκθεση αυτή. Είναι πολύ καλό η Επιτροπή, οι πολίτες να αναφέρονται στην Επιτροπή Αναφορών, να απευθύνονται σε εμά, διότι είναι ένα στοιχείο της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Δηλαδή, αν έχουν κάποια παράπονα, οι πολίτες είναι πολύ σκόπιμο να μπορούν να αναφερθούν στην Επιτροπή μας και αναφέρομαι και εγώ στο παράδειγμα Τη προστασία των ισπανικών ακτών, διότι οι πολίτες απευθύνονται σε μας για θέματα όπου η Κομισιόν αμφισβητεί την αρμοδιότητά μας. Όμως εμείς ε, κάνουμε το διάλογο με τους πολίτες, καθώς και με τα κράτη-μέλη, και σε ορισμένες περιπτώσεις ε, επιτυγχάνουμε αλλαγές υπέρ των πολιτών. Είναι λοιπόν μια κατάσταση όπου κερδίζουν όλοι, διότι διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να έχουμε συνομιλητές. Δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπο της ευρωπαϊκής ε, οικοδόμησης και αποδεικνύει και στους πολίτες ότι εμείς ως ε, ευρωπαϊκοί ευρωπαίοι πολιτικοί όντως ε, δεν περιοριζόμαστε σε γραπτές απαντήσεις. Κάτι μένει. Η Ισπανία λοιπόν είναι ένα παράδειγμα όπου και οι πολίτες αλλά και η χώρα και η Επιτροπή μας επέτυχε ουσιώδη πράγματα. Κάτι που θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε επίκαιρο στην ε, έκθεσή μας. Πρέπει και εμείς ε, στη διοίκησή μας να καταστήσουμε σαφές ότι έχουμε μια κάποια ειδική ε, θέση ως Επιτροπή Αναφορών. Είμαστε για τους πολίτες, δεν είναι οι πολίτες για μας. Εάν λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να συζητήσουμε ένα θέμα, εάν πιστεύουμε ότι το πρόβλημα πρέπει να το εξετάσουμε και επιτόπου, Δεν μπορούμε να περιμένουμε να εγκρίνονται οι επισκέψεις μας αυτές μέσω της κανονικής γραφειοκρατικής διαδικασίας. Δεν το καταλαβαίνουν οι πολίτες ε, αυτό. Πρέπει να είμαστε σε θέση να πάμε να διαπιστώσουμε την κατάσταση επιτόπου. Πρέπει να το κάνουμε σύντομα. Γιατί υπάρχει θέμα κατανόησης ε, με τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε την συνηθισμένη διαδικασία. Οι δικές μας ε, αντιπροσωπείες που κάνουν επιτόπου ε, αποστολές είναι μικρές, είναι ευέλικτες. Δεν είναι δυνατόν να μας λένε από τώρα να μας πείτε τι αποστολές θα κάνετε του χρόνου. Τα προβλήματα δεν μπορεί να τα προβλέψει όλα κανείς, προκύπτουν. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα διότι η ιστορία με τις ε, αποστολές fact-finding δεν έχει διευκολυνθεί, αντίθετα έχει γίνει πιο περίπλοκη και δημιουργούμε προβλήματα στον εαυτό μας. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Τσίτσιστερ. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους όπως είπα και για τη συνεργασία τους. Ένα θέμα που δεν ανέφερα στην εισαγωγή μου, ενώ θα έπρεπε, είναι τα διάφορα θέματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Ισπανία και τον νόμο για την παράκτια ζώνη. Θα προσπαθήσω βέβαια να είμαι αρκετά συνοπτικός για το θέμα αυτό για να μην φαίνεται ότι καταναλώνουμε μόνο γι' αυτό, είναι σημαντικό θέμα, αλλά δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι μας έχει γίνει έμονη ιδέα. Αυτό είναι ένα τμήμα της ε, εργασίας που θα κάνουμε για συμβαστικές τροπολογίες. Θα συναντηθούμε σήμερα το απόγευμα. Α, και θέλει ο κύριος Κάσμα να μιλήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Τσίτσεστερ που θέλησε να μου δώσει το λόγο με αυτό που συνήθως αποκαλεί διαδικασία Βουλής των Κοινοτήτων. Ίσως να μην ξέρετε όλοι ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού κάνει μια αποστολή fact-finding στην Ισπανία σήμερα. Θα πρέπει να καταλάβουν πόση δουλειά έχει κάνει η Επιτροπή μας ε, όχι μόνο μέσω των προηγούμενων τέτοιων αποστολών αλλά και μέσω των συστάσεων που έχει κάνει θα μπορούσατε ίσως ε, να το συμπεριλάβετε στην έκθεσή σας, στις επισκέψεις που κάναμε και που θα γίνουν τώρα. Χαιρόμαστε για αυτή την επίσκεψη. Λοιπόν, ε, αναλαμβάνω την Προεδρία, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Θέλει να πει τίποτα περαιτέρω ο εισηγητής. Όχι ή μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση. Εντάξει, τα είπατε όλα. Ωραία. Όλα σαφή. Ωραία. Να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογίων 12 Ιουλίου Οπότε όλες οι ομάδες παρακαλούνται να υποβάλουν τροπολογίες. Ε, οι σκιώδες ηγητές και ο συγητής ε, περιμένουν τις τροπολογίες ο κύριος Τσίτσεστερ. Θα ψηφίσουμε στις 12 Ιουλίου. Θα ψηφίσουμε στις 12 Ιουλίου. Νομίζω ότι έχει ήδη κλείσει η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Γι' αυτό έχουμε 110. Ε, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ε, ήθελα να δω αν προσέχει ο εισηγητής αυτά που λέω. Γι' αυτό τα είπα ε, αυτά. Ωραία. Η ψηφοφορία, όπως αναφέρει η Μέρση Δένταξη, θα γίνει στις 12 Ιουλίου. Ωραία. Και τώρα έχουμε το σημείο 9, τροπολογία για τον ε, προπολογισμό, ε, προσανατολισμό 2013, εισηγητή ο κύριο Σαλαβράκο. Οπότε του δίνω το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Επιτροπή μας αναλαμβάνει τη σύνταξη της γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013. Η γνωμοδότησή μου κινείται στο ίδιο ύφο με τα προηγούμενα χρόνια και συντάχθηκε με βάση την κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το οικονομικό έτος 2013, την οποία υπέβαλε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με το άρθρο 31. Τα μόνα σημεία που θα ήθελα να επισημάνω είναι αυτά που αφορούν την αύξηση του φετινού προϋπολογισμού κατά 3,89% και η οποία αύξηση αφορά τεχνικούς λόγους. Βασικά η αύξηση ενοικίου στο Στρασβούργο, καθώς η αναγκαστική μετακίνηση των γραφείων σε καινούρια γραφεία στις Βρυξέλλες, καθίσταται απαραίτητη αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να μετατρέψει τα γραφεία του Μεσολαβητή σε μουσείο. Συνεπώς δεν πρέπει να ε, επιρρύψουμε σε αυτό κάποια ιδιαίτερη υπέρβαση του προϋπολογισμού διότι η μετακίνηση καθίσταται αναγκαία και συνεπάγεται αύξηση του κόστους εν καιρό ε, βεβαίως κρίσης για το Κοινοβούλιο. Βεβαίως όσον αφορά την αύξηση των πιστώσεων για συμβασιούχους κατά 113.000 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες που μου παρασχέθησαν, είναι απόλυτα φυσιολογική και υπόκειται στο Γενικό Κανονισμό του Προσωπικού. Αυτά είναι τα δύο βασικά σημεία, αγαπητοί συνάδελφοι, που θα ήθελα να σας αναφέρω για να μην προβληματιστείτε ιδιαίτερως για την αύξηση του μπάτζετ. Κυρίως εκεί οφείλεται. Και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, όπως και εγώ, θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και θα περιμένω με χαρά τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για να δω, θέλει κανείς το λόγο. Θέλει κανένα να συμπληρώσει, να προσθέσει κάτι. Δεν βλέπω. Ήταν η έκθεσή σας τόσο αναλυτική που είναι όλοι ευχαριστημένοι. Θαυμάσια. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε στις 12 Ιουλίου, έτσι αναφέρεται. Παρακαλώ να προετοιμαστείτε όλοι. Επόμενο θέμα, το σημείο 10. Γνωμοδότηση για την έκθεση, για την εφαρμογή της Χάρτας ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Η συγγήτρια, η συνάδελφος Βάλεαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, κατά τα τελευταία χρόνια ένα τρίτο των αναφορών που έχει λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφορούσε ισχυριζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αναφέρεται στο χάρτη ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, η έκθεση Ιθαγένειας του 2010 όπως επίσης και η έκθεση προόδου προς την αποτελεσματική Ιθαγένεια ε, του 2010 συμπέραναν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν ασκούν τα δικαιώματα τη ηθαγένεια του, Οι προσδοκίε ε, των Ευρωπαίων πολιτών και διαμενόντων που ζητούν ε, την ε, καταγγελία της παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κάτι το οποίο αναφέρεται και στις συνθήκες και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι αποτέλεσμα της περιορισμένης ερμηνείας της, ε, του, του ρόλου ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή των σχετικών νόμων. 48% των αναφορών ισχυρίζονται ότι δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι οι πολίτες για τα δικαιώματά τους και είναι ένα από τα βασικά εμπόδια στην διασυνοριακή κυκλοφορία και παρεμποδίζει την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών ήθελα να συζητήσω ορισμένε από τι παραβιάσει των θεμελιωδών δικαιωμάτων που εντοπίσαμε και στην έκθεσή μα και ε, που κατά τη γνώμη μας ε, πρέπει να ε, αποκατασταθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Πρώτα απ' όλα το, η δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων, των επαγγελματικών προσόντων, της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και των, ε, ε, της ασφαλιστικής κάλυψης είναι πάρα πολύ σημαντικά σε σχέση με την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όμως πολλοί ε, αναφέρουν ότι οι πολίτες έχουν πρόβλημα με την εξασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα αυτά την χάνουν σεβασμού ε, εφαρμογής ε, και ανάπτυξη. Υπάρχει ένα νομικό κενό σε σχέση με ε, την αποζημίωση όταν ε, τα κράτη-μέλη καθυστερούν στη μεταγραφή της ε, νομοθεσίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει ότι όχι μόνο μεταγράφεται η νομοθεσία αυτή από τα κράτη-μέλη αλλά ότι γίνεται σωστή εφαρμογή των νόμων προκειμένου να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών πολιτών. Προτείνουμε λοιπόν ε, η σχετική έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα να συμπεριλαμβάνουν την αξιολόγηση εφαρμογή ηθαγένεια στα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, γίνει, να κάνει μία ε, ετήσια διάσκεψη από κοινού με, με την Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ ε, για να υπάρξει συζήτηση των εμπλεκομένων φορέων για το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει επιγόντως ε, ότι η Οδηγία 38 ε, του 2004 όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εφαρμόζεται σωστά και το λέω αυτό σε σχέση με τις αναφορές που αφορούν τα προβλήματα μεταξύ άλλων νομίμως διαμενών των αλλοδαπών χωρών τρίτων χωρών, όπως επίσης και την κάλυψη των ε, συζύγων ή συντρόφων τους. Ε, υπάρχει επίσης και το θέμα της ελευθερίας των μέσων μαζικής των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση του θέματος αυτούς και πρέπει να υπάρξει νομοθεσία ώστε κοινέ προδιαγραφές για τον πλωραλισμό των μέσων ενημέρωσης ε, όντως επιβάλλονται. Ένα ακόμη ευαίσθητο θέμα, αντικείμενο αναφορών που λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η κατάσχεση ε, ακίνητης περιουσίας ε, όταν ελεύθερα μετακινούνται σε κάποια χώρα τη ευρωπαϊκή Ένωση. και επίση ε, ζητώ στην έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανανεώσει τον ε, ε, κανονισμό για την ίδρυση του Οργανισμού Ανθρωπίνων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προκειμένου να ενισχύσει το ρόλο και την εξουσία του. Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω πρώτα απ' όλα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη γνώμη της. Ο κύριος Δεσμέτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την ε, εισηγήτρια. Να σας ε, πω ότι εμείς από την πλευρά της Κομισιόν συμφωνούμε με την ανάλυση ότι υπάρχουν υψηλές προσδοκίες από την πλευρά των πολιτών σε ό,τι αφορά τη χάρτα που τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 2009 και που έδωσε μία όθηση ε, στα πράγματα από τότε. Επίση, αυτό επιβεβαιώθηκε από μια πρόσφατη μελέτη που ζητήθηκε από την Κομισιόν, τα πόρισματα τη οποία μα έδειξαν ότι η γενική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χάρτα αυξήθηκε σημαντικά αλλά η ακριβής ε, γνώση ε, περί χάρτας είναι σχετικά χαμηλή. Αυτό επιβεβαιώνεται και από πολλές καταγγελίες που λαμβάνει η Επιτροπή κάθε χρόνο 3.260 καταγγελίες περίπου λάβουμε, 216 καταγγελίες λάβαμε το 2011. Έχουμε μια στρατηγική που ευθετήθηκε το 2010, μια στρατηγική σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή της χάρτας ε, και καθιστά προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορεί να κατηγορηθεί όταν νομοθετεί για θέματα που αφορούν ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αξιολογήσαμε την ε, προόδο για την εφαρμογή της στρατηγικής το 2011 στην ετήσια έκθεση του 2011 σχετικά με την εφαρμογή της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τι βλέπουμε ότι υπάρχει μια θετική τάση, δηλαδή γίνεται ένα σημείο αναφορά σε όλο και περισσότερο η χάρτα και για τα ευρωπαϊκά όργανα όταν νομοθετούν, αλλά και ε, για εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, ε, καθώς και για τα δικαστήρια, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, μια σειρά αποφάσεων του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου που αναφέρονται στη χάρτα και είδαμε ότι από το 2010 στο 2011 έχουμε περίπου 50% περισσότερες αποφάσεις ε, με αναφορά στη χάρτα, με παραπομπή στη χάρτα. Έτσι λοιπόν αυτή είναι σημαντική εξέλιξη και θα συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε τα επόμενα έτη. Επίση, η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη σέβονται τη χαρτά όταν εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο στην ε, ετήσια μας έκθεση ανακοινώσαμε ότι θα επιζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της χάρτας. Φυσικά οι ανησυχίε των πολιτών ε, είναι ένα κεντρικό ζήτημα για την Επιτροπή και θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες ε, για να βοηθήσουμε τους πολίτες ε, να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλίων όπως η δημοσίευση πληροφοριών ε, για την πύλη e-justice ηλεκτρονικής δικαιοσύνης Επίσης, ε, για τους μηχανισμούς ε, προσφυγής ε, σε εθνικό επίπεδο σχετικά με παραβίαση, περίπτωση παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων και επίσης θα συνεχίσουμε το έργο μας και θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε, ενθαρρύνοντας, παραδείγματος χάρη, καταγγελίες όπως στο Διαμεσολαβητή και σε άλλους οργανισμούς για να έχουμε ένα checklist παραδεκτού, έτσι ώστε να διευκολύνουμε και την προσφυγή σε ένδικα μέσα και να βοηθήσουμε τους πολίτες ε, να κατανοήσουν αν οι καταγγελίες τους ε, μπορούν να είναι αντικείμενο διαχείρισης από, τον αρμόδιο, από το φορέα που έχουν στείλει τις, όπου έχουν στείλει τις καταγγελίες. Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που τίθενται από την συγκέντρωση, όπως ε, παραδείγματος χάρη, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τα τρία ευρωπαϊκά όργανα μπορούν να ζητήσουν ε, γνωμοδοτήσεις από τον ε, Οργανισμό Θεμελιωτών Δικαιωμάτων για συγκεκριμένα ζητήματα και σε ό,τι αφορά την ε, τροποποίηση του κανονισμού Έχουμε μία εξωτερική αξιολόγηση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή για τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συνεχίζεται το έργο αυτό και θα υπάρξει και παρακολούθηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί αυτό το έργο πριν να εξετάσουμε Τώρα θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον κανονισμό. Και τέλος, να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να ακολουθεί μία ε, εντατική πολιτική σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών. Ευχαριστώ. Να αναφέρω το προφανές ότι θέλουμε μια θαυμάσια παρουσίαση στο ίντερνετ για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μπορείτε να τη δείτε στο ίντερνετ. Γιατί είπαμε ότι ορισμένε φορέ υπάρχουν προβλήματα επικοινωνία, πολλοί πολίτε δεν ξέρουν καν τα δικαιώματά του. Είναι πολύ καλό να υπάρχει δυνατότητα αυτή, οι πολίτες δηλαδή, να έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να βρουν εύκολα τα δικαιώματά τους. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η συζήτηση που γίνεται με βάση τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Πρέπει να γίνει η συζήτηση αυτή. Ε, ο μιλήτρια πρώτο, ο κύριο Μπάγκου. Και μετά ο κύριο Μπαστινάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σωστά τονίσατε αυτό που και εγώ ήθελα να τονίσω ως επιθυμία μου. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Βαλεάν για τη θαυμάσια εργασία την οποία επετέλεσε, όπου για μένα τουλάχιστον καθιστά σαφές ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά. Και είναι υποχρέωσή μας να τηρούνται, να μπορούν να ασκηθούν χωρίς δισταγμούς από κανένα κράτος μέλος ή από κανένα θεσμικό όργανο. Το σχέδιο γνωμοδότησης υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι ένα από τα πιο γνήσια όργανα που διευκρινίζει κατά πόσον γίνονται σεβαστά και ασκούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να τονίσω ότι για να ασκούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει ε, να υπάρχει ταυτόσιμη κατάσταση δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Ο... Η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν είναι κάτι που προέκυψε λόγω μικροπολιτικών συμφερόντων, αλλά είναι η βάση για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν πρέπει να έχουν τα θεμελιώδη δικαιώματα την ίδια έννοια, το ίδιο περιεχόμενο, τον ίδιο τρόπο άσκησης σε κάθε κράτος μέλος. Και οι κυρώσεις επίσης για μη σεβασμό πρέπει να είναι ταυτόσιμες. Γι' αυτό καλό για να εγκριθούν οι αναγκαίες τροπολογίες που θα το, διαβεβαιώσουν, θα το εξασφαλίσουν αυτό και συγχαίρω και πάλι την κυρία Βάλνα για την εργασία της. Ο συνάδελφος Μπαστινάρου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. επικροτώ την έκθεση αυτή. Πραγματικά είναι ένα ζήτημα πολύ επίκαιρο, όχι μόνο για την Επιτροπή Αναφορών, αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικά για, τους για τα ευρωπαϊκά όργανα, ειδικότερα όταν ε, υπάρχει κρίση και βλέπουμε πολύ συχνά τα κράτη-μέλη να νομίζουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα έρχονται δεύτερα και δεν είναι προτεραιότητα όπως θα έπρεπε να είναι η κανονική συμπεριφορά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, πρέπει να αξιολογήσουμε την ε, εφαρμογή ε, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εγώ διαφωνώ με αυτό που συχνά έχει επαναλάβει ε, η Επίτροπος ε, και ε, Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ όταν λέει ότι είναι οριζόντιο θέμα αυτό στην ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι αν θέλουν τα κράτη-μέλη μπορούν να το κάνουν καλώς, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Όχι, δεν γίνεται εμεί να κάνουμε μάθημα στην Κίνα, στη Ρωσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να βλέπουμε ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να υπάρχουν επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και να σιωπούμε ή να παραμένουμε αδρανείς. Επίσης, υπάρχει πολύ χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινού σε σχέση με την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την υποχρέωση των κρατών μελών να εφαρμόζουν σωστά το χάρτη αυτό και να ε, αξιοποιούν τις διατάξεις του και σε επίπεδο ε, πολιτών ε, με καλή, με παρκές επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης η ευαισθητοποίηση είναι πολύ χαμηλή, πολύ μικρή. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε, κάπως να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση για την εφαρμογή θεμελιωδών δικαιωμάτων, γιατί για την ώρα δεν είναι επαρκής. Υπάρχει και έλλειψη βούλησης ε, για την εφαρμογή από τα κράτη, ε, από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην σας πω ότι υπάρχουν και μερικά τα οποία θέλουν να φύγουν ε, από την σύμβαση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και μερικά κράτη-μέλη ακόμη αντιδρούν και δεν θέλουν να την εφαρμόσουν σωστά και αυτό είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο τα δύο τελευταία χρόνια βλέπουμε περιπτώσεις ε, ε, συμπεριφοράς κρατών μελών που κατάφορα παραβιάζουν ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Υπάρχουν νόμοι εθνικοί που, που στις διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, αντιδράσει ε, εκ των υστέρων όμως και προσπαθώντας απλώς να αποκαταστήσει μια ε, κατάσταση και δημιουργώντας διαφωνίες και συγκρούσεις που θα ήταν πολύ καλύτερο να τις είχαμε διαχειριστεί σε πρώιμο στάδιο όταν είχαμε δει ότι υπήρχε κίνδυνος να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ε, με την επίδοση ε, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, στην, στη Βιέννη και δεν φταίει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ κάνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Αντιπρόοδο, Αντιπρόεδρο και Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ να δείξει, να καταστήσει πιο ορατό και πιο ε, ουσιώδη τον οργανισμό αυτό. Πρέπει να έχει λίγο μεγαλύτερη σημασία η ύπαρξή του. Γιατί μιλάμε για ένα πολύ ζοβαρό ζήτημα, που είναι η εφαρμογή ε, του χάρτη θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων. Δεν είναι δυνατόν να έχει ένα δευτερεύοντα ρόλο απλώς στην όλη προσπάθεια που κάνουμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μια τελική παρατήρηση θα ήθελα να κάνω τα κριτήρια της Κοπεχάγης λέμε ότι είναι μόνο για την περίοδο την προενταξιακή. Και μετά τέλος, δεν κάνουμε τίποτα. Αν τα κράτη-μέλη δηλαδή καταφέρουν να μας πείσουν ε, ότι ε, τα καταφέρνουν επαρκώς για να μπουν ε, στην Ευρωζώνη, μετά δεν το ξεχνάνε εντελώ. Και από νομικής απόψεως αυτό το πράγμα είναι εντελώς αντιφατικό. Να μην σας πω ότι από ηθικής και πολιτικής απόψεως είναι απαράδεκτο. Διότι όταν ένα κράτος μέλος έχει προσχωρήσει προχωρήσει σε σε μια νομοθεσία είναι υποχρεωμένο να, να συμπεριφέρεται ε, στο πλαίσιο της νομοθεσίας αυτής. Αλλά μας έχει πει η Επίτροπος πολλές φορές «Α, όχι, αυτό είναι μόνο για τους αρχάριους, για αυτούς που θέλουν να προσχωρήσουν. Οι επόλοιποι είναι ήδη ε, όριμοι και δεν χρειάζεται να ε, τους ελέγχουμε» το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο στη δική μας ε, διάσκεψη της Επιτροπής Αναφορών μας είπε ότι ναι, είναι δεσμευτικά τα κριτήρια της Κοπενχάγης για τα κράτη-μέλη. Για ποιο ε, λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τόσο διστακτική στο να αποδεχθεί αυτό το πράγμα, ότι ένα νομοθέτημα πρέπει να είναι δεσμευτικό για τα κράτη-μέλη από τη στιγμή που θέλει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τη ε, στιγμή ε, που θέλει να φύγει. Ότι δεν είναι δυνατόν να ε, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους η εφαρμογή των ε, νόμων αυτών. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για το κοινό, γιατί από αυτά τα προβλήματα προκύπτουν ε, διάφορα προβλήματα κοινωνικής, οικονομικής φύσεως, ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, ελευθερίας των μειονοτήτων και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να τα λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό ακριβώς επικροτώ την προσέγγιση της ε, συναδέλφου Βαλέαν και είμαι πεπισμένος ότι θα ε, κλονίσει λίγο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έκθεσή μας για να ασχοληθεί με τα θεμελιώδη δικαιώματα σαν να είναι ένα ουσιώδες ζήτημα και όχι ένα θέμα που το συζητάμε που και που όταν υπάρχει μια κρίση γιατί χωρίς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά θα υπάρξουν νέες κρίσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βίκτορ. Γέλνα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω λοιπόν όσα ήδη αναφέρθηκαν για τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι πολύ βασικό έγγραφο, είναι τμήμα της Εθνικής Λισαβόνας, είναι λοιπόν ε, ένα από τα πιο σημαντικά νομοθετήματα γενικά του ευρωπαϊκού δικαίου. Και γι' αυτό Χαίρομαι με τη γνωμοδότηση. Θα καταδείξει εάν και κατά πόσο και με ποιο τρόπο γίνεται σεβαστή χάρτα σε κάθε κράτος μέλος. Ωστόσο, να αναφέρω ακόμη ότι υπάρχουν δύο χώρες από τις 27, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είναι νομικά δεσμευτική χάρτα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να οθήσουμε αυτές τις χώρες να εισαχθεί στο δίκαιό τους η χώρα, ε, στο δίκαιό τους η χάρτα. Θα προτείνω λοιπόν μια τροπολογία σε αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Η κυρία Όκεν. Δεν θέλω να επιμηκύνω τη συζήτηση. Υποστηρίζω τον Σάνφο Μπαστινάρου για την ανάγκη να είμαστε πολύ πιο σαφείς. Διότι πολύ συχνά η Κομισιόν διστάζει να ασχοληθεί με βασικά θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κάναμε μια ακρόαση όπου πολλοί είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό και πρέπει οπωσδήποτε, μια που υπάρχει αυτή η υπηρεσία, Όλοι θέλαμε να υπάρξει αυτός ο νέος φορέας, αλλά ορισμένοι ισχυροί δεν θέλουν να υποστηριχθεί η εργασία της. Υποστηρίζω λοιπόν την εργασία αυτού του οργανισμού. Ευχαριστώ. Βεβαίως θα δώσω το λόγο και στην εισηγήτρια, αλλά έγιναν πολλές προτάσεις. Ο Βίκτορ αναφέρθηκε σε πολύ σημαντικά θέματα το ένα είναι γενικό. Ορισμένες φορές η Επιτροπή είναι κάπως ε, αφελής. Όταν υπάρχουν ε, νομοθετήματα που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα, ε, θεωρεί δεδομένο η Κομισιόν ότι θα τα εφαρμόσει το, το, τα κράτη-μέλη. Θα τα μεταγράψουν στο τεχνικό τους δίκαιο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη. Πρέπει να ελέγχουμε εάν όντως υπάρχει αυτή η εφαρμογή. Επειδή όμως αυτή η διαδικασία είναι ένας μαραθώνιος, όταν ε, προσπαθεί να ενταχθεί μια χώρα στην Ένωση, όταν λύγει αυτός ο μαραθώνιος, όταν μπαίνουν στην Ένωση, τότε λένε ωραία δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε την προσπάθεια, μπορούμε να χαλαρώσουμε. Εμείς ως Επιτροπή Αναφορών διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αναφορές των πολιτών, διαμαρτυρίες για μη εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή για άνηση από κράτος σε κράτος. Πρέπει να υπογραμμίσουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εισηγήτρια. Θα διαπίστωσε η εισηγήτρια ότι σε στηρίζουμε και σας δίνω το λόγο για το κλείσμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για όλα τα σχόλιά τους. Ε, σας ευχαριστώ και για το πόσο παθιασμένοι είστε με το θέμα και νομίζω δικαίως. Σε σχέση με αυτό το ζωτικό θέμα για μας ε, ως πολίτες της Ένωσης. Και πράγματι πιστεύω ότι είναι ένα θέμα επί του οποίου θα είμαστε ενωμένοι παραδοσιακά η Επιτροπή μας υποστήριζε, δηλαδή να ε, προσπαθεί το Κοινοβούλιο να είναι προοδευτικό και να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα διασφαλίσω ότι και για αυτό το θέμα θα ισχύει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα σχόλιά σας και τη συνεισφορά σας στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία για την έκθεση αυτή θα γίνει στις 12 Ιουλίου. Σωστό? Ωραία. Έχουμε λοιπόν αρκετές ψηφοφορίες ε, τον Ιούλιο. Πολλή εργασία πρέπει να επιτελεστεί μέχρι τότε. Επόμενο θέμα. Αναφορά ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα είναι αναφορές κατά της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση των απομιμήσεων, άκτα, με 2,8 εκατομμύρια υπογραφές, ε, δεν το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό, οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε αρμόδια επί της ουσίας επιτροπής, επιτροπή, αλλά είμαστε μια επιτροπή που ασχολείται με τα αιτήματα των ε, πολιτών Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να μας απασχολήσει αυτή η αναφορά. Σήμερα λοιπόν για πρώτη φορά προσπαθούμε να συζητήσουμε αναλυτικά το θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Άλεξ που εκπροσωπεί μέσω της παρουσίασής του επιθυμεί να εκπροσωπήσει 2,8 εκατομμύρια ελπίζω να επιτύχει αυτή την εκπροσώπηση και μετά θα μιλήσει και ο David Μάρτιν και μετά η Κομισιόν. Αλλά πρώτα απ' όλα από πλευράς ε, των αναφερόντων ο κυριο Άλεξ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδιαίτερη ικανοποίηση για μένα να βρίσκομαι εδώ και προσωπώντας 2,8 εκατομμύρια ανθρώπου στην Επιτροπή Αναφορών προκειμένου να εκπροσωπήσω τη μεγάλη ανησυχία που αισθάνονται πολλοί πολίτες για τη Συμφωνία Άκτα. Όταν έχουμε σύγκρουση δικαιωμάτων δεν θα πρέπει οι πολίτες να είναι σαν θεατές σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, δηλαδή απλώς να είναι θεατές και να μην μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα όταν διακυβεύονται οι ελευθερίε μα θα πρέπει να υπάρξει μια δέουσα διαδικασία για να διασφαλίσουμε ότι γίνονται σεβαστές οι ελευθερίε μα και ότι ενισχύονται. Η ΑΚΤΑ, η Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση τη παραποίηση, ε, είναι ακριβώ το αντίθετο. Η διαπραγμάτευση έγινε και κλεισμένων των θυρών και θα καθιστούσε ένα νομικό καθεστώ όπου οι ιδιωτικέ εταιρείε ε, δεν θα λογοδοτούν και ουσιαστικά θα παρακολουθούν το διαδίκτυο. Κάποια στιγμή όταν ε, άνθρωποι κατεπεσμένοι στη Μέση Ανατολή διαγυνδέμουν τη ζωή τους για να κερδίσουν την ελευθερία τους, οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πήραν τα στυλό τους ε, για να καταργήσουν κάποιες από αυτές τις ελευθερίες, καθώς έδειξαν πολύ μεγάλη ανησυχία για να προστατεύσουν πραγματικά πνευματικά τους δικαιώματα. Υποστήριξε ομάδες όπως η DRA είναι ε, η ε, αρμόδια υπηρεσία για τα ψηφιακά δικαιώματα. Πολίτες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μας προσέγγισαν και απευθύνθηκαν σε μας για να αναλάβουμε δράση. Η αβάς ε, που σημαίνει σε πολλές γλώσσες φωνή ή τραγούδι είναι ένα νέο είδος κινήματος ε, των πολιτών. Πιστεύουμε ότι είναι το μεγαλύτερο κίνημα των πολιτών που ενεργοποιεί πολίτες σε διεθνή θέματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και απαντήσαμε με μία αίτηση η οποία ε, έριξε ε, ευρύ φως όλη την Ευρώπη και πέρα της Ευρώπης και τώρα έχει υπογραφεί, όπως είπε και ο Πρόεδρος, από πάνω από 2,8 εκατομμύρια ανθρώπους. 2,84 εκατομμύρια άνθρωποι υπέγραψαν πρόσφατα τους τελευταίους μήνες αυτή την αίτηση, αυτή την αναφορά. Και λέει, και απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ό,τι αφορά του παγκόσμιου πολίτε, σα καλούμε να υπερασπίσετε ένα ανοιχτό και ελεύθερο διαδίκτυο και να απορρίψετε την κύρωση ε, τη εμπορική συμφωνία κατά τη παραποίηση τη ΑΚΤΑ που δεν το κατέστρεφε. Το διαδίκτυο είναι ένα ζωτικό εργαλείο για ανθρώπου σε όλο τον κόσμο να ανταλλάσσουν ιδέε και να προωθούν τη δημοκρατία πρέπει να δείξουμε πραγματική παγκόσμια ηγεσία γιατί και θες και να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας οι διαπραγματευτές της ΑΚΤΑ ακολούθησαν τη λανθασμένη διαδικασία και εκπώνησαν λανθασμένη συμφωνία με λανθασμένο συνόλο χωρών και λανθασμένους μηχανισμούς επιβολής. Αλλά μαζί ε, πολίτες που επιγραμμούμε και ε, βουλευτές με τις κατάλληλες αρμοδιότητες μπορούν να πετύχουν το κατάλληλο αποτέλεσμα, δηλαδή να απορριφθεί η άκτα. Αν δούμε τι έγινε το 2000, αν δουν τι έγινε το 2012, μελλοντικοί ιστορικοί μπορούν να δουν τώρα την απόφαση που επίκειται να λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ως ε, μια προστασία ε, των πολιτών και υπέρ της λογοδοσίας ε, επιμένει ε, πολίτες ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει το λέγειν όταν διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση διεθνεί συνθήκε. Εδώ εκπροσωπώ σήμερα του πολίτε που καλωσορίζουν ε, τι αποφάσει ε, των τριών επιτροπών αυτού του Κοινοβουλίου που συστήνουν να απορριφθεί η άκτα. Τώρα, η, Διεθνής, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου αυτή την εβδομάδα καλείται να αποφασίσει και καλούμαστε να ακολουθήσουμε και να απορρίψουμε την άκτα και στην Ολομέλεια αυτού του Κοινοβουλίου επίσης πρέπει να γίνει το κατάλληλο βήμα, το υπεύθυνο βήμα και να μην συνενέσει επί της κύρωσης και να διασφαλίσει ότι η συμφωνία αυτή δεν θα δει ποτέ το φως της μέρας. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτή την Επιτροπή, την Επιτροπή Αναφορών, για τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο της, ε, καθώς βοήθησε να διοχετευτεί φωνή των πολιτών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 2,8 εκατομμύριων πολιτών εδώ, σε όσου λαμβάνουν αποφάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στα υπόλοιπα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να έχουμε τέτοιε επιτροπέ και διάβλου που θα διασφαλίζουν ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθεται να συζητήσει διεθνεί συμφωνίε, ότι θα θέτουν πρώτα τι θεμελιώδει ελευθερίε και θεμελιώδη δικαιώματα και δεν θα τα παζαρεύουν έναντι οποιοδήποτε εμπορικού συμφέροντο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτήν την σύντομη και περιεκτική παρουσίαση. Οπότε θα δώσω για μια σύντομη τοποθέτηση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος λόγή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος θα πάρει το λόγο? Ευχαριστώ. Η Επιτροπή ε, έχει πλήρη συνείδηση των ανησυχιών των πολιτών και κάποιων μη κυβερνητικών οργανισμών για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια της ΑΚΤΑ. Επανειλημμένα έχουμε επιχειρήσει να καθησυχάσουμε τις ανησυχίες αυτές διότι η άκτα κυρίως στοχεύει στη βελτίωση του σεβασμού των ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας παγκόσμια και γύρω σε τρίτες χώρες. Η άκτα δεν εφαρμόζεται απευθείας στους Ευρωπαίους πολίτες. Και ακόμη πιο σημαντικό, η άκτα δεν τροποποιεί την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και ούτε άμεσα ούτε έμεσα δεν παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης όπως αναφέρονται στη χάρτα. Επανειλημμένα το έχουμε αναφέρει, η νομική υπηρεσία και του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν δώσει διαβεβαιώσεις από αυτού. Η άκτα εξετάζεται από τους νομομαθείς, από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, σε όλα τα κράτη-μέλη και με ομόφωνη στήριξη των κρατών μελών τελικά η Ένωση αποφάσισε να υπογράψει αυτή την συμφωνία. Αλλά επειδή παραμένουν αμφιβολίε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να ζητήσει την τελειωτική γνώμη για τέτοιου τύπου θέμα έκανε έτοιμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ούτω ώστε να δώσει την οριστική γνωμοδότηση για την συμβατότητα της άκτα με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και έχουμε κάθε εμπιστοσύνη ότι αυτή η γνωμοδότηση θα επιβεβαιώσει τη δική μας εκτίμηση. Γιατί έχουμε εντολή να διαπραγματευτούμε, ξέρουμε ότι μια διεθνή συνθήκη δεν μπορεί να παραβιάζεται να θέτει ένα αμφιβόλο ενωσιακά δικαιώματα και έχουμε εμπιστοσύνη γιατί αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα αναφέρονται σαφώς στην συνθήκη άκτα, στο γράμμα της. Αναφέρθηκαν κάποια προβλήματα με το διαδίκτυο. Αλλά το άρθρο για το ίντερνετ, την άκτα, είναι ένα μόνο. Αναφέρεται εκπεφρασμένα στην ανάγκη προστασίας της ελευθερίας του λόγου, της ιδιωτικής σφαίρας, της προστασίας των δεδομένων. Αναφέρονται λοιπόν και προστατεύονται στο κείμενο. Δεν πρόκειται να παραβιαστούν. Ακούμε τη φωνή των πολιτών, προσπαθούμε να διευκρινίσουμε, να είμαστε απόλυτα σαφείς Ελπίζουμε το δικαστήριο θα ε, διευκρινίσει τελειωτικά το θέμα και θα ήταν σκόπιμο να λεφθεί υπόψη και άψη του δικαστηρίου λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία γιατί μιλήσατε για την σωστή διαδικασία που πρέπει να υιοθετηθεί για την ε, έγκριση αυτής της συμφωνίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να ακουστεί και το δικαστήριο και είναι επίσης πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει γιατί είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα των εταιριών της για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης, φυσικά πάντοτε σεβόμενοι τα, θεμελιώδη και ουσιώδη δικαιώματα, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι έχουμε επιτύχει αυτό το στόχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν να ε, ανοίξω τώρα το κατάλογο μιλτών, να σε ενημερώσω ότι η πρώτη αναφορά ε, για την άκτα ελήφθη από την ΠΕΤΗ το 11. Διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου έχουν ήδη συζητήσει για την άκτα και την έχουν απορρίψει η Επιτροπή Ανάπτυξης, Βιομηχανίας, η ΛΥΜΠΕ και η Νομική Επιτροπή και σήμερα ε, οργανώσαμε αυτή τη συζήτηση γιατί την Πέμπτη η ΙΝΤΑ που είναι αρμόδια επί της ουσίας ως ε, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα συζητήσει το θέμα αυτό και η Επιτροπή θα λάβει υπόψη και τη γνώμη των αναφερόντων και των άλλων εισηγητών και ο εισηγητής της ΙΝΤΑ, ο Ντέβιτ Μάρτιν που είναι παρόν οπότε θα προτιμούσα να του δώσω πρώτο το λόγο. Κύριε Μάρτιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή που με προσκάλεσε. Ευχαριστώ τον Άλεξ και τους υπόλοιπους αναφέροντες ε, για την ενεργό συμμετοχή τους ε, στην όλη συζήτηση επί της άκτα. Όταν η ε, με έχρισε ε, η εισηγητή. Ελπίζω να έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση. Ε, πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι πολίτες ήταν πάρα πολύ ενεργοί ε, στο να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους στους ευρωβουλευτές. Ε, το επικροτώ αυτό, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα ε, οι πολίτες ήταν έτοιμοι να συνεργαστούν ενεργά με ευρωβουλευτές, όχι μόνο μέσω υπογραφής μιας αναφοράς, αλλά με ε, αποστολή ε, email προκειμένου να συμμετέχουν στη συζήτηση και εμείς δεν πρέπει να αρκεστούμε απλώς στο να τους απαντάμε στα γράμματά τους. Η άποψή μου έρχεται κάπως καθυστερημένα, αλλά ούτως ε, ή άλλως ε, ε, οι ίδιοι οι πολίτες ε, οι ίδιοι οι δημιουργοί ε, συμμετείχαν στην όλη διαδικασία. Όταν δεν έχουν πολύ μεγάλο εισόδημα και βλέπουν και εκείνοι ότι η άκτα δεν είναι η κατάλληλη συμφωνία, πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη κάτι τέτοιο. Και αυτό το επικροτώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, δυνάμει βέβαια όλων όσων συνέβησαν για τη διαπραγμάτευση της ΑΚΤΑ έχουν ε, και εκείνοι συμμετάσχει πολύ ενεργά, ήρθαν σε πολλές συνεδριάσεις και στις διαπραγματεύσεις αλλά και στις συζητήσεις ε, και προσπάθησαν να την υπερασπιστούν. Έξι κοινοβουλευτικές ε, επιτροπές ε, θα έχουν ε, συζητήσει μέχρι το τέλος της διαδικασίας αυτής. Τέσσερις έχουν διαφωνήσει και η πέμπτη θα ψηφίσει την πέμπτη οι αναφέροντες ελπίζω να καταλάβουν συνεπώς ότι έχουμε πάρει σοβαρά το θέμα αυτό, ότι το έχουμε συζητήσει πολύ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα ε, υπό διάφορε οπτικές γωνίες, αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, στο διεθνές εμπόριο, στις ελευθερίες του πολίτη, ε, στις ε, υπόλοιπε διαδικασίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να μπω σε πάρα πολλέ λεπτομέρειες όσον αφορά το περιεχόμενο σήμερα, το έχω κάνει πολλές φορές άλλωστε. Θα ήθελα απλώ να πω ότι αν δεν είχαμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, δεν θα είχαμε την άκτα. Και κατά πόσο είναι, το, το, και του αν κάποιος είναι υπέρ ή κατά της άκτα, το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η φωνή των πολιτών σημαίνει ότι μπορεί να εξετάσει λεπτομερώς το ζήτημα και να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα και αυτό πρέπει να ε, θεωρείται ευπρόσδεκτο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα ε, και ε, ήταν αντικείμενο ανοιχτή ε, εξέταση από όλου. Και το βλέπω από το τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Βουλή των Κοινοτήτων έχει ένα σύστημα βάσει του οποίου κάποιοι μπορεί να προτείνουν τη συζήτηση ενό θέματος όταν θεωρούν ότι είναι διαφιλονικούμενο. Η άκτα είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά αυτόν τον τρόπο και ε, η ενεργό συμμετοχή των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως είπα και προηγουμένως. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Άλεξ ήταν τόσο ε, δραστήριος στην όλη διαδικασία, όπως και οι υπόλοιποι συμπολίτε του και θα ήθελα και εκείνο να τον ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ανοίγουμε τον κατάλογο μελετών. Πρώτος ο συνάδελφος Μάφη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας ε, της ΓΚΟΕ θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους αναφέροντες όχι μόνο όσου υπέγραψαν ε, την αίτηση, ε, αλλά όσου συμμετείχαν και στι διαμαρτυρίε ε, σε όλη την Ευρώπη και μάλιστα σε πολλέ περιπτώσει είχαμε μεγάλε διαμαρτυρίε. Πρέπει να του ευχαριστήσουμε και να του εχαρούμε, γιατί χάρη στην κινητοποίηση των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη έχουμε μια σοβαρή συζήτηση σήμερα σε αυτό το κοινοβούλιο για το θέμα τη ΑΚΤΑ και γι' αυτό ίσως ε, μπορεί να σημειώσουμε μια μεγάλη νίκη και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την άκτα. Κατά την άποψή μου αυτό οφείλεται μόνο στην πίεση που ήρθε μαζικά εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η δική μου πολιτική ομάδα ήταν κατά της άκτα από την αρχή και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και όταν θα συζητηθεί το θέμα στην Ολομάλη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την άποψή μου ουσιαστικά κράτησε μια λαζονική στάση στη συζήτηση αυτή και προσπάθησε απλώς ε, να ψηφίσει την όλη αντίθεση που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη λέγοντας ε, ότι ε, έχουν παραπληροφορηθεί οι άνθρωποι και δεν γνωρίζουν γιατί πράγμα μιλάμε όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ μίλησα με πάρα πολλούς από όσους συμμετέχουν στην εκστρατεία και εγώ πιστεύω ότι η Κομισιόν κάνει αυτό που κάνει συνήθως η Κομισιόν δηλαδή υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ευρώπη έτσι λοιπόν για αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις επιχειρήσεις ε, προέρχεται ε, η άκτα από το λόμπι που άσκησαν ε, τα μεγάλα εμπορικά επιμελητήρια και θέτουν τα κέρδη πάνω από τα βασικά δικαιώματα των πολιτών και αν δούμε και πώ έγιναν οι διαπραγματεύσει, ε, ε, βλέπουμε ότι υπάρχει περισσότερο διαδικτύου, μετατρέπονται σε αστυνομικού. Επίση υπάρχουν επιθέσει ε, κατά τη πρόσβαση στα γενώσιμα φάρμακα. Αλλά νομίζω ότι εδώ είμαστε στο χείλο τη νίκη, είμαστε στα πρόθυρα τη νίκη και θα ήθελα να ενθαρρύνω όσοι συμμετέχουν στην εκστρατεία να συνεχίσουν να ασκούν πίεση. Αν μπορούσαμε να ασκήσουμε πίεση και τελικά τα καταφέρουμε στην ΙΝΤΑ, θα μπορέσουμε να να τα καταφέρουμε και στην Ολομέλεια. Και ουσιαστικά αυτό θα είναι το αποτέλεσμα μια μαζική εκστρατεία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι 8 έχουν ζητήσει το λόγο. Οπότε θα πρέπει να μιλήσω καθένας ε, γύρω στα τρία λεπτά γιατί θέλουμε και ο αναφέρον να μπορέσει να πάρει το λόγο στο τέλος ε, για να εφαρμόσουμε λοιπόν τη σωστή διαδικασία. Λοιπόν σας παρακαλώ γύρω στα τρία λεπτά παρακαλώ Εντάξει, παρακαλώ, Ντέβιτ, να μου πεις ε, όταν ε, θα έχουν παρέλθει τρία λεπτά. Η κυρία Τσουάν Λόκα και μετά η κυρία Μιράντα. Εγώ είμαι. Ευχαριστώ. Έχω ήδη ως μέλος της ΛΥΜΠΕ και της ομάδας μου που εκπροσωπείται εδώ εκφράσει την άποψή μου και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και όλοι είμαστε κατά της άκτα και υπέρ της αρνητικής άποψης της ε, ΛΥΜΠΕ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, αναφέροντες τόσο μεγάλος αριθμός ατόμων. Επειδή προέρχομαι από την Λετωνία, θέλω επίσης να αναφέρω που, ότι, είναι η πρώτη, ότι η πρώτη αναφορά για το θέμα αυτό το 2011 προέκυψε από Λετωνό πολίτη. Οι πολίτες της Λετωνίας δεν έχουν αποστείλει πολλές αναφορές, αλλά ήμασταν πρώτοι για το θέμα αυτό. Βεβαίως οι επικριτές μας λένε ότι δεν έχουμε ενημερωθεί σωστά. Αλλά ένα παράδειγμα από τη Λετωνία καταρρύπτει τους χειρισμούς τους. Την προηγούμενη εβδομάδα ο βοηθός μου συμμετείχε σε μια συζήτηση στο ραδιόφωνο με εκπροσώπους της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου Βεβαίως οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης ήταν υπέρ της Άκτα αλλά κατάφερε να αποδείξει ότι δεν είχαν καν διαβάσει τα κύρια σημεία της έκθεσης και δεν είχαν καμία εμπιστοσύνη στα επιχειρήματά τους ενώ τα δικά μας είναι πολύ ισχυρά και χαίρομαι που για το θέμα αυτό το Κοινοβούλιο συμφωνεί με τις απόψεις των αναφερόντων. Τα μικρόφωνα δεν δουλεύουν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συνάδελφος η κυρία Βελιέ ε, ασχολείται πάρα πολύ με, το, αυτό, αλλά δεν μπορεί σήμερα να βρεθεί εδώ γιατί εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Σύνοδο Κορφή στο Ρίο. Μου ανέθεσε λοιπόν εξ ε, της ε, ομάδας ε, των Πρασίνων ε, να σας αναφέρω το εξή σήμερα στο ιστορικό της Επιτροπής μας εξετάζουμε την αναφορά κατά της άκτα. Ε, πρόκειται για μια αναφορά που υπεγράφει σχεδόν από 3 εκατομμύρια άτομα. Πρόκειται ε, με, για τον ίδιο πληθυσμό που έχει και η πατρίδα μου, η Γαλλικία. Τρία εκατομμύρια άτομα και ε, ουσιαστικά είναι τρεις φορές περισσότερο, μεγαλύτερος ο αριθμός των πολιτών που έχουμε για την πρωτοβουλία των πολιτών. Και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με αυτή τη Διεθνή Συμφωνία αυτό το ζήτημα πρέπει να ενισχύσει τις δικές μας ε, ευθύνη. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να ψηφίσει επί της άκτα τον Ιούλιο. Σήμερα τέσσερις κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, ήδη κάλεσαν να απορριφθεί η συμφωνία αυτή. Να απορριφθεί και οι συνάδελφοί μας ε, ως ε, υπογράφοντες της αίτηση αυτής ε, θεώρησαν ότι δεν σέβεται η συμφωνία αυτή τα θεμελιώδη δικαιώματα προστατεύονται από τη Χάρτη των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων έτσι λοιπόν αυτές οι επιλές είναι πραγματικές. Ε, ο Ευρωπαίος Υποπτής ε, Προστασίας των Δεδομένων ε, και ο ίδιος είπε ότι οι διατάξεις της ΑΚΤΑ θα μπορούσαν να σημαίνουν παρακολούθηση των πολιτών στο διαδίκτυο online και η συμφωνία αυτή παραβιάζει την προστασία των δεδομένων και της προσωπικής ζωής στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο βάσει της νομολογίας το επέμενε στο ότι η παρακολούθηση δεν μπορεί να είναι ε, γενική και έτσι λοιπόν η άκτα δεν ε, εγγυάται κάτι τέτοιο. Γι' αυτούς λοιπόν τους λόγους ε, και οι συνάδελφοι μου και εγώ ζητώ εξ ονόματος της ομάδας αλλά και εξ ονόματος των, της Ευρώπης να εγγυηθούμε τα προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών ε, που μας εμπιστεύονται το καθήκον αυτών ε, και να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή και ε, προκειμένου να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα για την Ευρώπη, ένα ισχυρό μήνυμα, δηλαδή θέλουμε να δώσουμε φωνή στους πολίτες. Äh, Ευχαριστώ. Κυρία Γέλνια Και μετά κυρία Ρόμενα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους σήμερα μπορούμε να συζητήσουμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής μας αυτήν την αναφορά που μας υπενθυμίζει ότι για λόγους που δεν καταλαβαίνω καθυστέρησε ένα μήνα. Τέλος πάντων σήμερα συνεδριάζουμε, τη συζητούμε. Η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με την κατάσταση το 2009 γιατί τότε αρχίσαμε να ε, σας ενημερώνουμε για τις απειλές ε, που προέκυπταν από την άκτα Είχαμε τότε, είχε χαθεί και ένα ψήφισμα της δικής μας ομάδας σε σχέση με τον αντίκτυπο, σε σχέση με, την, ε, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης όταν άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Έπρεπε να είχαμε ε, συμπεριλάβει το θέμα αυτό και να είχαμε συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και βάση περιπτώσει μετά εμφανίστηκε αυτή η συμφωνία μέσα από πολύ περίεργες διαδικασίες διαδικασίες. Υπήρξαν όμω φωνέ στο Κοινοβούλιο κατά τη συμφωνία αυτής και επιτέλους ε, όταν ο κόσμος βγήκε στους δρόμους ε, κάποιοι βουλευτές επιτέλους διάβασαν το κείμενο ε, και ξύπνησαν. Ξύπνησαν επιτέλους. Επειδή λοιπόν ε, με πολύ δημοκρατικό τρόπο οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους και ε, χάρη στους, στις αναφορές, ε, χάρη στο ότι μπορούν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτοί το ίντερνετ μπορούμε να διαφωνήσουμε σήμερα με την άκτα. Υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία κατά τη άκτα στο ε, Κοινοβούλιο, όμως δεν είναι πάρα πολύ σαφές ακόμη και στην τελευταία επιτροπή που θα συζητηθεί το θέμα αυτό την Πέμπτη, ελπίζω η άκτα να πάψει να υπάρχει μια για πάντα και ελπίζω και στην Ολομέλεια να συμβεί αυτό. Όσον αφορά τώρα στη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το, Φεβρουάριο είπε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα απέστειλε το κείμενο στο ε, δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Περίμεναν, μετά είπαν ότι το ξανάστηλαν και ότι περίμεναν ε, την απάντηση. Επιτέλους το Μάιο έλαβαν ε, τα ε, σχετικά στοιχεία, κάτι το οποίο βέβαια καθυστέρησε πάρα πολύ ολόκληρη την ε, διαδικασία και αναγκαστήκαμε και εμείς να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Εμείς είχαμε αναλύσει ούτως ή άλλως λεπτομερώς το κείμενο. Είναι ένα επικίνδυνο κείμενο. Ε, θέλουμε χρηστή νομοθεσία και αυτή η νομοθεσία δεν κειμενο θελουμε χρηστη χρηστή. Η κυρία η κυρια Α, με συγχωρείτε. συγχωρείτε ο κύριος Ρωμέρα Ιρουέβα. Εγώ θα επιμείνω σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, όχι στους λόγους γενικά για τους οποίους πρέπει να διαφωνήσουμε με την ΑΚΤΑ. Δεν είναι μόνο θέμα μιας συζήτηση για την ομοθεσία, είναι μια πολιτική συζήτηση και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τεθεί. Δεν συζητούμε μόνο το περιεχόμενο του κειμένου αυτού, συζητάμε στην ουσία πώς αυτό το κείμενο προέκυψε, που είναι το πιο σημαντικό ζήτημα, και δεύτερον, ποιες θα είναι οι συνέπειες του κειμένου αυτού αν εγκριθεί με τον τρόπο με τον οποίο έχει προταθεί ω τώρα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική και η αναφορά αυτή. Είναι τόσο σημαντικό ε, που ε, εκατομμύρια ε, πολίτες θίγονται και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να αυξήσουμε την αξιοπιστία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αν δεν κάνουμε αυτό που αναμένεται από εμά, από εμάς τους ε, εκλεγμένους ε, εκπροσώπους, θα χάσουμε τέλος πάντων τη λίγη ε, αξιοπιστία που μας ε, έχει μείνει. Γι' αυτό δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία αυτή. Όσοι συνάδελφοι δεν το έχουν κατανοήσει ακόμη αυτό, παρακαλώ κατανοήστε το. Δεν είναι μόνο ένα νομικό ζήτημα, ένα ζήτημα που έχει να κάνει μόνο με το νομικό κείμενο. Θα χάσουμε την ευκαιρία να ε, αυξήσουμε την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμών. Ωραία, ε, ωραία. Πρώτα απ' όλα η κυρία Κέλλα και μετά ο κύριος Μπαστινάρο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς ε, και τους ε, 2,8 εκατομμύρια πολίτε ε, που υπέγραψαν την αίτηση αυτή και φαίνεται πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για αυτό το ζήτημα. δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε πανευρωπαϊκά κινήματα όταν υπάρχουν ε, ζητήματα που κινητοποιούν του πολίτε σε όλη την Ευρώπη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη αυτέ τι αναφορέ, Αλλά όχι μόνο να τι λαμβάνουμε υπόψη αλλά και να λαμβάνουμε και δράση. Θα ήθελα να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα θυγούν από την άκτα που δεν έχουν ε, τη δυνατότητα να καταθέτουν ε, αναφορές, κυρίως άνθρωποι σε άλλες χώρες, κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες που θα υποφέρουν ε, από τους κανονισμούς περί και έτσι λοιπόν θα υπάρχει δυσχερής πρόσβαση στα γενώσιμα φάρμακα και θα αναρωτηθείτε τι έχει να κάνει η ΑΚΤΑ, αλλά ε, περιορίζοντας ε, θέματα εμπορίου σε ό,τι αφορά τα εμπορικά σήματα, μπορεί να υπάρχουν πολύ σημαντικές συνέπειες ε, για τη ζωή και την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων. Όμως οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να καταθέτουν αναφορές, δεν μπορούν να έλθουν εδώ στο Κοινοβούλιο, όμως πάντοτε πρέπει να τους έχουμε κατά νου όταν συζητούμε τέτοια θέματα, πρέπει να δίνουμε και σε άλλους ανθρώπους τη δυνατότητα να υψώσουν τη φωνή τους εδώ, γιατί η ΑΚΤΑ μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή τους. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την αναφορά και ελπίζουμε να έχουμε και ορθή έκβαση, μια αίσια έκβαση στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Ευχαριστώ, Μπαστινάρο. Και να προετοιμάζεται η κυρία Όκεν. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω την αναφορά και εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών χαιρόμαι πάρα πολύ που δηλώνω ότι η δική μας πρόταση να θεωρηθεί ως ε, κατεπήγον θέμα η άκτα για την Επιτροπή Αναφορών έγινε ε, δεκτή από το Προεδρό και από τους συντονιστές. Τώρα συζητάμε αυτό το θέμα και είναι ζωτικό. Τώρα, για το περιεχόμενο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό που προκλεί το δικό μου ενδιαφέρον και όχι μόνο το δικό μου ενδιαφέρον, μας είπαν ότι πρόκειται για ένα καλό μέσο για να αντιμετωπίσουμε την παραποίηση κτλ. Αλλά αυτό που είναι τόσο προφανές είναι Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τα μέσα για να προστατεύσει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Γιατί στα υφιστάμενα μέσα να προσθέσουμε και κάτι άλλο, γιατί να μην βελτιώσουμε όσα υπάρχουν σήμερα αντί να δεκτούμε την άκτα. Κατόπιν μα είπαν αυτό είναι ένας τρόπος ε, για την κατεπολέμηση των παροπημένων προϊόντων. Είναι απαράδεκτο γιατί οι κύριοι παραγωγοί και τους καλοπαραγωγούς, τους αποκαλοπαραγωγούς των παραποιημένων αγαθών δεν είναι αυτοί που θα ε, δεσμεύονται από αυτή τη συμφωνία. Δεν υπάρχει ούτε μία λέξη για όσους παράγουν αυτά τα αγαθά. Έτσι λοιπόν καταπολεμούμε την παραπίστηση στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι σοβαρό κάτι για την πολιτική διάσταση τη ιδέα αυτή. Εμεσούσει τη κρίση. Οπότε ε, υπάρχει και αφαίρεση κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα, οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάζει αυτή την ιδέα να δημιουργήσει μια αστυνομία του διαδικτύου. Αυτή είναι η μόνη δημοκρατική απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Δηλαδή πολιτικά είναι εντελώς λάθος. Δεν είναι μόνο απαράδεκτο, αλλά πρέπει και να την απορρίψουμε. Και εδώ καλωσορίζω την άποψη που παρουσιάστηκε από πολλούς πρωθυπουργούς στην Ευρώπη, από την Πολωνία μέχρι και τη Ρουμανία, τη δική μου χώρα. Αν όλοι είμαστε ενωμένοι στο να καταγγείλουμε και να απορρίψουμε την άκτα, τότε σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και αν ένα μεγάλο μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη δήλωσε ότι είναι αντίθετο στην άκτα. Και αναφέρομαι και στη δική μου ομάδα των σοσιαλιστών σήμερα. Αν τόσες πολλές επιτροπές ήδη δήλωσαν ότι δεν είναι αποδεκτή η συμφωνία αυτή και θα έπρεπε να απορριφθεί και την απέρριψαν. Μπορούμε να δαπανούμε το χρόνο μας σήμερα και να λέμε στο τα στείλουμε στο δικαστήριο και να δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Και κατόπιν να το εκτούμε. Όχι, όχι. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το χρόνο, πρέπει στο Κοινοβούλιο μαζικά να καταψηφίσουμε την άκτα και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Κοιτάξτε, προσπαθώ εδώ να περιοριστώ. Να τα πω έτσι, δεν είναι καλό για το κύριο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι καλή η συμφωνία αυτή για την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού μα μοντέλου. Το αντίθετο. Ουσιαστικά καταστρέφει την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού μοντέλου στα μάτια εκατομμυρίων ε, πολιτών στην Ευρώπη, αλλά όχι και μόνο. Και εδώ δεν συζητάμε μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα μοντέλο που επιτρέπει παγκόσμια έφοδο και πώς θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες. Δεν πρέπει να περιορίζουμε την πρόσβαση στην ελεύθερη πληροφορία, ούτε πρέπει να περιστέλουμε τις ελευθερίες. Έτσι λοιπόν υποστηρίζω πλήρως την αίτηση αυτή, την αναφορά αυτή και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει μαζική ε, απόρριψη τσάκτα από αυτή την Επιτροπή καταρχήν και κατόπιν θα ακολουθήσει και η Ολομέλεια. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Κυρία Άουκεν. Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να αρκεστώ στα τρία λεπτά. Μπορεί όμω να είμαι και συντομότερη. Νομίζω ότι θα πρέπει να γιορτάζουμε σήμερα. Να γιορτάζουμε το γεγονό ότι φαίνεται επιτέλου το αποτέλεσμα τη συνθήκη τη Λισαβόνα, ε, ότι έχει ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν, είμαστε, δεν είναι απλώ κάποιο με τον οποίο ε, πρέπει να είμαστε καλοί και να κάνουμε διάλογο. Γίνεται συναπόφαση πλέον και θα ήταν πολύ καλό αν οι, τα άλλα δύο όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το καταλάβουν αυτό μια και καλή για να μην αλλαχάνουμε και το χρόνο μας. θα έπρεπε να ρωτήσουμε όντως και το δικαστήριο ποια είναι η άποψή του για το κείμενο αυτό και κατά πόσο ευσταθεί νομικά. Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των αναφερόντων, των πολιτών και των ε, εκπροσώπων τους στο Κοινοβούλιο. Θα, μπορούσαμε, θα μπορούσαν ε, ε, να μας πούνε όχι, μην, ξο... μην ε, χάνετε χρόνο ούτε χρήματα πηγαίνοντας στο δικαστήριο γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Έχουμε προβλήματα λοιπόν με την αξιοπιστία μας και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να γιορτάζουμε. Τον Ιούλιο θα δείξουμε ότι οι πολίτες ε, εκλέγουν ένα κοινοβούλιο το οποίο διαδραματίζει το ρόλο του. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Γιάρα. Όχι, ο κύριος Βίλαντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω από την αρχή τη συζήτηση γιατί ήμουν στην ΑΦΚΟ όπου ε, παρουσίασα ένα θέμα ε, που αφορά τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να δημιουργεί εξεταστικές επιτροπές όπου ακριβώ τίθεται το θέμα. Έχουμε το δικαίωμα αυτό και πώς θα το ασκούμε ως κοινοβούλιο. Επ' αυτού ε, το Συμβούλιο ε, έχει κάποιες αντιρρήσεις. Όμως θα ήθελα να νερώσω λίγο το κρασί μας. Υπάρχουν πράγματα που τα αντιμετωπίζουμε εμείς με έναν τρόπο και που ξαφνικά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο. Διότι έχει αρχίσει ήδη να επισέρχεται και το στοιχείο της ε, προεκλογικής εκστρατείας. Όταν βλέπω εδώ, για παράδειγμα, αυτά τα μπλουζάκια που έχετε βάλει, αυτό θεωρώ πως δεν είναι σωστή κοινοβουλευτική πρακτική. Δεν θέλω ούτε διάφορα άλλα πανιά, ούτε σημαίες εθνικές να βλέπω. Οι βουλευτές έχουν άλλες δυνατότητες να εκφραστούν. Είναι ιδιαίτερα επίμαχο το θέμα αυτό. Το θέμα αυτό εκρεμεί, είναι σκόπιμο. Όταν τα θέματα εκρεμούν και έχουν ε, και νομική πλευρά, να μην τα αντιμετωπίζουμε. Γιατί εμείς, ε, ε, μιλάμε, εμείς συζητάμε ε, για θέματα όπου έχουν εξαντληθεί τα νομικά μέσα. Υπάρχουν πολλοί ζωτική σημασία θέματα όπου λέμε θέλουμε να ακούσουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος ή της, της Συνταγματικής Επιτροπής και τώρα που γίνονται όλες αυτές οι συζητήσεις στο σώμα, εμείς προσπαθούμε να προτρέξουμε. να αμφισβητήσιμο αυτό. Θα πρέπει να αφήσουμε τις υπεύθυνε και αρμόδιες επί να κάνουν αυτό που κάνουμε και εμείς για τα δικά μας θέματα. Να αφήσουμε τις επί της επιτροπές να, κάνουμε, να κάνουν τη δουλειά τους. Ανήκω σε αυτήν την επιτροπή από τότε που εξελέγει προβουλευτή. Και πάντα δεν είναι σαφές αν είναι σωστό να στηρίξουμε ή να απορρίψουμε κάποιο θέμα. Πάντα προσπάθησα να δημιουργήσω μια υπόλοιψη αντικειμενικής αντιμετώπισης των θεμάτων. Και για μένα, ανεξάρτητα από το πώς υπογράφουν μια αναφορά ένας ή πολλοί, δεν έχουμε βρει ακόμη το σημείο όπου το γεγονός ότι κάποιοι υπογράφουν μία αναφορά αν είναι την καθιστά ορθή. Αν κάποιος υπογράψει μόνος του μία αναφορά και την υποβάλει ακόμη και αν είναι ένας εάν η Επιτροπή μας θεωρεί σωστή την αναφορά πρέπει να το στηρίξουμε. Δεν έχει να κάνει με το αν έχει υπογραφεί μία αναφορά από έναν ή από εκατομμύρια. Υπάρχει η δυνατότητα αιτήματο ε, δημοψηφίσματος αν υπογράψουν πολλοί. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να εξετάσουμε αυτήν την αναφορά με τη συνηθισμένη διαδικασία. Διότι αν κάνουμε λάθος ε, μπορούμε να αλλάξουμε και άποψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ε, κατάλαβα ακριβώς ε, τι είπε ο κύριος Βίλαντ. Φαίνεται ότι πιστεύει πως η δική μας Επιτροπή δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και θα έπρεπε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε άλλες επιτροπές. Όμως εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι σχεδόν 3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες εξέφρασαν τη θέση τους ε, για το θέμα αυτό. Ναι, πράγματι υπάρχει και η πρωτοβουλία των πολιτών, ε, δυνάμει τη συνθήκη της Λισαβόνας και αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Όμως, εδώ έχουμε τρία εκατομμύρια πολίτες ε, που υπέγραψαν μία αίτηση και πρέπει να τους χαρούμε. Και πάνω από τέσσερις επιτροπές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψαν τη συμφωνία αυτή και παραμένει μόνο η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου να τοποθετηθεί. Και τέλος, οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μας πιστεύουν ότι αυτό το θέμα δεν είναι μόνο νομικής φύσεως, αλλά πιστεύουν ότι και εμείς ε, ως εκπρόσωποι των πολιτών θα έπρεπε να τοποθετηθούμε. Είναι πολιτικό ζήτημα και το γνωρίζετε πολύ καλά. Όποια και είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εμείς ε, εδώ εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Ευχαριστώ. Τέιλορ. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει κάτι να πω για να υποστηρίξω τους συναδέλφους μου. Υποστηρίζω ιδιαίτερα και έντονα αυτές τις αναφορές που μας καλούν να μην επικυρώσουμε την άκτα. Και χαίρομαι που ήδη τέσσερις επιτροπές του Κοινοβουλίου μας έχουν κάνει ακριβώς αυτό. Φυσικά πιστεύω ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στην Επιτροπή Αναφορών, ακόμη και αν είναι μόνο ένας ή δύο ή χίλιοι. Είναι καθήκον μας να τους εξηγήσουμε πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο, να ανταποκριθούμε στο αίτημά τους. Αλλά δεν είναι μόνο μερικοί. Και επίσης ε, τέσσερις επιτροπές συναδέλφων μας είπαν ότι θέλουν να απορριφθεί εντελώς η άκτα. Υποστηρίζω λοιπόν τις ε, προτάσεις που έχουν γίνει η Επιτροπή μας να καλέσει την Ίντα Βεβαίω θα πάρει θέση μόνη της, αλλά να λάβει υπόψη ότι οι συνάδελφοί τους πολλών επιτροπών έχουν ήδη αποφασίσει να απορριφθεί η άκτα διότι η άκτα θα έχει αρνητική επίδραση στο ε, δίκαιο εμπόριο, στην διαδικασία ψηφιοποίησης και στην διοίκηση του ίντερνετ και σε άλλους τομείς. Θέλουμε να υποστηρίξουμε λοιπόν ε, αυτές τις αρνητικές επιδράσεις. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε την ε, δραστηριότητα. Συμφωνώ λοιπόν με τους αναφέροντες. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η τελευταία παρέμβαση. Τώρα θα δίνω το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Βίλξ για να απαντήσει σε σχέση με τα σχόλια που ακούστηκαν. Σας ευχαριστώ. Όταν ε, ήρθε εδώ στις αρχές Μαΐου εντυπωσιάστηκα με το καλωσόρισμα της Επιτροπής ε, Αναφορών και τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης μετέφεραν ε, την ευρωπαϊκή φωνή μακριά και πραγματικά με εντυπωσίασε το πώς διαχειρίστηκε αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν ασχολήθηκαν μόνο μία-δύο επιτροπές με αυτό το θέμα αλλά έξι επιτροπές και νομίζω ότι σήμερα είναι πολύ σημαντική ημέρα και πετύχαμε μία συμφωνία ε, η οποία ήταν, διαπραγματεύτηκε ε, μυστικά και ε, ουσιαστικά κάποιες ε, εταιρείες να παρακολουθούν τα άτομα στο διαδίκτυο. Ουσιαστικά καταφέσαμε να ρίξουμε φως σε αυτή τη συμφωνία και φυσικά όλο αυτό σημαίνει ότι τώρα δεν είναι πρακτικά δυνατόν να υπογραφεί στις επόμενε δύο εβδομάδε. Καλούμε την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και κατόπιν την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου να μην περιμένει, αλλά τι επόμενε δύο εβδομάδε να κάνει το αποφασιστικό βήμα απόρριψη τη άκτα, γιατί είναι λανθασμένη αυτή η συμφωνία, η διαπραγμάτευση έγινε με λανθασμένο τρόπο και έτσι πραγματικά πρέπει να απορριφθεί, πρέπει να ακουστεί η φωνή των πολιτών. Και χαίρομαι και που η Άβας διαδραμάτισε ένα ρόλο στο να διοχετεύσει το θυμό ε, και τις ανησυχίες των μελών μας στην Ευρώπη και ελπίζω να κάνει το καθήκον του το Κοινοβούλιο και να διασφαλίσει ότι η άκτα δεν θα τεθεί εφαρμογή και οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία που θα διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακούσει και τη φωνή των πολιτών και των Ευρωπαίων Βουλευτών από την αρχή της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ. Ε, εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιάρμο έχει ζητήσει το λόγο για να καταθέσει μια πρόταση. Ευχαριστώ επειδή είχα προεδρεύσει και λιγάκι, να κάνω μια διαδικαστική πρόταση και να μιλήσω στην Επιτροπή. Φυσικά δεν είμαστε πολιτική επιτροπή, αλλά δεν είμαστε και επί της ουσίας για το θέμα αυτό. Είμαστε η Επιτροπή Αναφορών. Πολλές επιτροπές έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό, έξι συγκεκριμένα. Αλλά συνήθως εμείς ως Επιτροπή Αναφορών συνεργαζόμαστε στενά με τις επί της ουσίας αρμόδιες. Αυτονόητο. Υπάρχει και μία προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, προτείνω να κρατήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά για να μπορούν και οι αναφέροντες ε, να υποβάλουν νέα στοιχεία και ως συνήθως θα συνεχίσουμε να συζητάμε και να διαπραγματευόμαστε για το θέμα αυτό. Να την κρατήσουμε λοιπόν ανοιχτή αυτή την αναφορά. Θα περιμένουμε τις απόψεις των άλλων επιτροπών και θα αποφασίσουμε κατόπιν διότι αφορά πολλούς τομείς αυτή η έκθεση ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αναφέροντες για την κοινή τους ενέργεια αλλά εφόσον η επί της ουσίας Επιτροπή ε, δεν θα, η, θα συζητήσει το θέμα και δεν θα τη συζητήσουμε εμείς επί της ουσίας θα θέλουμε να ακούσουμε την άποψη και των άλλων επιτροπών. Να κρατήσουμε λοιπόν ανοιχτή την επιτροπή και να συνεχίσουμε να συζητάμε και να καθορίσουμε από κοινού τη διαδικασία με τις αρμόδιες της ουσίας επιτροπές. Παστινάρο. Ευχαριστώ. Βεβαίω, είμαι υπέρ να την κρατήσουμε ανοιχτή. Αλλά το ερώτημά μου είναι ανοιχτή γιατί τέσσερι επιτροπές έχουν ήδη λάβει θέση. Είναι κατά τη άκτα. Βεβαίω, να την κρατήσουμε ανοιχτή αλλά ποια είναι η θέση μας για το περιεχόμενο της άκτα. Είμαστε υπέρ του να την κρατήσουμε απλώς ανοιχτή ή ναι, την κρατάμε ανοιχτή αλλά η Επιτροπή μας να δηλώσει ότι είναι κατά της άκτα. Αυτή την ε, πρόταση τροπολογίας κάνω. Αυτό μας δίνει την αξιοπιστία αλλά και τη συμμετοχή. Να την κρατήσουμε ανοιχτή δεν ισχύει. Μπορούμε να ενώσουμε τη φωνή μας με τις τέσσερις φωνές επιτροπών που εκφράστηκαν σαφώς κατά. Μάρτιν. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι επισκέπτης, δεν θα μιλήσω για το τελευταίο σημείο, αλλά έχει σημαντικό ρόλο η Επιτροπή Αναφορών. Μετά την άκτα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά ας υποθέσουμε ότι η ΙΝΤΑ θα πει όχι και ότι η Ολομέλεια θα πει όχι αλλά εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπόθεση. Δεν ξέρω αν το δικαστήριο θα συνεχίσει τη διαδικασία εξέταση του θέματο αν απορρίψει το Κοινοβούλιο την άκτα, αλλά αν το κάνει, τότε η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να συζητηθεί κάπου στο δικαστήριο. Και επειδή υπάρχει αυτή η αναφορά ενώπιον τη Επιτροπή σα, θα μπορούσατε εσεί να είστε λογικό χώρο για να συζητηθεί. Διότι δεν ξέρω εάν θα ήταν σκόπιμο να πάει στην Επιτροπή ΙΝΤΑ πρέπει να δώσετε μία ε, απάντηση στις ανησυχίες του αναφέροντος. Ίσως λοιπόν θα ήταν η κατάλληλη επιτροπή εδώ να συζητηθεί από του δικαστηρίου. Θα μπορούσε να έρθει ενώπιόν σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Μάρτιν ε, για τη συμμετοχή του. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες. Ευχαριστώ και τον κύριο Βίλξ ε, που μας παρουσίασε και μας υποστήριξε την αναφορά αυτή. Εγώ πιστεύω ότι μία πρώτη απάντηση στο αίτημα που προήλθε από τον κύριο Μποστινάρου δόθηκε από την καταληκτική παρέμβαση του εκπροσώπου των ε, πολιτών που υπέγραψαν. Αυτή είναι μια σημαντική ημέρα γιατί υλοποιήθηκε ουσιαστικά το καθήκον της Επιτροπής μας. Δηλαδή ουσιαστικά να δίνεται δυνατότητα στους πολίτες να ασκούν πλήρως το δικαίωμα της θεγενειάς τους και αυτό συνέβη και να δίνουμε προβολή όχι μόνο στην Επιτροπή αλλά και στο ζήτημα που θεωρούν πάρα πολύ ε, σημαντικό τόσοι πολίτες. Έτσι λοιπόν, ε, να, ε, το να λέμε εδώ ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια που δεν μπορεί να γνωριθεί. Και αυτό μου επιτρέπει να απαντήσω και στο υπόθηκαν από τον κύριο Βίλαν. Ε, δεν είναι ο μεγάλος αριθμός ε, που μας οθεί στο να εξετάσουμε μία αναφορά ε, και να τη θέσουμε πάνω από μία άλλη. Γιατί κάθε φορά ξέρουμε ότι ακόμη και ένας πολίτης να καταθέσει μία αναφορά θα πρέπει να συζητηθεί αυτή στην Επιτροπή μας. Είναι σαφές ότι υπάρχει υπάρχει μια διαφορετική πρόθεση από τη στιγμή που είναι τόσοι οι πολίτες, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διευρυμένη δυσαρέσκεια και πρέπει να δράσουμε πιο γρήγορα σε σχέση με άλλες υποθέσεις. Όμως την ίδια προσοχή δίνουμε όλες τις αναφορές η συζήτηση που έγινε και ε, νομίζω ότι οι περισσότεροι ε, ουσιαστικά θέλουν να λάβει θέση αυτή η Επιτροπή γιατί νομίζω ότι πάνω από 12 συνάδελφοι τοποθετήθηκαν και όλοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους ε, σε σχέση με αυτή την υπόθεση της υπογραφής της συμφωνίας. Η δική μας διαδικασία βέβαια προβλέπει να μην λαμβάνεται απόφαση επί της ουσίας, αλλά να παρακολουθούμε ε, την αναφορά των πολιτών. Έτσι λοιπόν, ε, τώρα για το ερώτημα του κ. Μποστινάρου, τι θα κάνουμε εμείς. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να απαντήσουμε ως εξή. Με την πρόταση του συναδέλφου Γιάρ. Να αφήσουμε βεβαίως ανοιχτή την αναφορά, και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, πώς εξελίσσεται το ζήτημα στις ε, αρμόδιες επιτροπές ε, και ε, στο Κοινοβούλιο και ενώπιον του δικαστηρίου. Και κατόπιν η Επιτροπή μας αφήνοντα πάντοτε ανοιχτή την αναφορά, θα αποτελεί ένα έσχατο μέσο προσφυγής για τους πολίτες, εκεί όπου αυτές οι διαδικασίες δεν θα ανταποκρίνονται στα συμφέροντα των πολιτών. Αν οι συνάδελφοι λοιπόν συμφωνούν με την ανάλυση μου και με το συμπέρασμα αυτό, θα έλεγα εγώ να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και φυσικά ε, συμπεριλαμβάνουμε και τα πολιτικά σχόλια που ακούστηκαν στη συζήτηση, θα παρακολουθούμε ε, πώς ε, θα εξελιχθεί το ζήτημα στις υπόλοιπες επιτροπές αλλά και στο δικαστήριο και θα ξαναπροτείνουμε μια συζήτηση για να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις, έτσι λοιπόν. Ολοκληρώνουμε εδώ τη συζήτηση για αυτή την αναφορά, η οποία παραμένει ανοιχτή για μελλοντικέ αποφάσει από την Επιτροπή μα. Ευχαριστούμε του αναφέροντε και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος, έκανα λάθο. Όχι, έκανα λάθο. Νομίζω ότι τα είχαμε αναβάλει όλα, αλλά έχουμε το σημείο 12 έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο. για την έκθεση αυτή ε, που αρμόδια της οποίας ήταν η κυρία Γιώτοβα που ήταν και επικεφαλής της αντιπροσωπείας θα δώσω λοιπόν το λόγο στη συνάδελφο για να μας πει ποιε δραστηριότητες πρέπει εμείς να αναλάβουμε στα πλαίσια των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήδη σας είχα πει ορισμένα πράγματα για την αποστολή μας στο Βερολίνο. Βασίστηκε σε απόφαση της ε, Επιτροπής μας και ήταν επίσης και αποτέλεσμα πολλών καταγγελιών και αναφορών ε, σε σχέση με το ρόλο των ε, υπηρεσιών νεολαίας Jugendamt. Jugendamt. Στις 4 Μαΐου υπήρξε σχετικό κείμενο, ε, υπήρξε, έγινε πολλή δουλειά προκειμένου να υπάρξει ε, συνένεση κατόπιν συζήτησης. Πήγαμε λοιπόν στο Βερολίνο, κατόπιν καταγγελιών ε, ότι η Jugendamt ε, παραβιάζει τα δικαιώματα των παιδιών. Εμείς δεν πήγαμε εκεί να κατηγορήσουμε κανέναν, ε, πήγαμε εκεί γιατί θέλαμε να προτείνουμε μια επικοδομητική λύση. Βεβαίως δεν θέλουμε να παρέμβουμε στα εσωτερικά μιας χώρας, αλλά ε, υπάρχει προφανώς ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την επικοινωνία, υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης ε, ε, για το δικαστικό σύστημα, δεν υπάρχει διάλογος και αυτό καταλήγει βεβαίως σε παρεξηγήσεις αλλά και σε δικονομικά προβλήματα. Τι γίνεται σε περίπτωση πληροφοριών ε, όταν ε, υπάρχει ένα διασυνοριακό διαζύγιο. Πολλές από τις καταγγελίες που έλαβε η Επιτροπή μας έλεγαν ότι οι ε, αλλοδαποί γονείς δεν μπορούσαν να μιλούν στα παιδιά τους στη γλώσσα τους ε, όταν υπάρχει κίνδυνος, ε, για παράδειγμα, απαγωγής του παιδιού. Όταν δεν υπάρχει διερμηνία ή όταν δεν μιλάει τη γλώσσα του γονιού ο υπάλληλος της Jugendamt. Παρόλα όλα αυτά, δεν θα έπρεπε να δημιουργείται πρόβλημα με αυτό το γλωσσικό θέμα θέμα, γιατί η γλώσσα είναι αυτή που δημιουργεί μια γέφυρα και θα έπρεπε όλες οι γλώσσες να μπορούν να χρησιμοποιούνται. Οι επαφές μεταξύ παιδιών και γονέων δεν θα έπρεπε να είναι περιορισμένες, θα έπρεπε να είναι τακτικές και να ενθαρρύνονται. Εμείς λοιπόν υποβάλαμε τις προτάσεις μας ε, βάσει των όσων διαπιστώσαμε και μετά συζητήσαμε με διάφορους εκπροσώπους ε, ε, άλλων οργανισμών. Ήταν βέβαια σύντομη η επίσκεψή μας και αποστήλαμε γραπτό ερωτηματολόγιο στις ε, σχετικές αρχές, λάβαμε εγγράφος απαντήσεις και αυτό μας βοήθησε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο ε, ζήτημα Γι' αυτό ε, ακριβώς ε, ήταν ε, μεγάλη προθεσμία για την εκπόνηση του εγγράφου. Θα έχετε κι εσείς περισσότερο χρόνο για να σκεφτείτε τις τροπολογίες και τις προτάσεις σας. Συζητήσαμε κατά πόσο οι προτάσεις θα μπορούσαν να γίνουν μόνο από τα μέλη της αποστολής, γιατί μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουν την καλύτερη πληροφόρηση αλλά σκεφτήκαμε μήπως θα μπορούσαμε να, προ... να επιτρέψουμε και σε άλλους συναδέλφους ε, να υποβάλουν συστάσεις βάσει των εγγράφων ε, ε, των συνοδευτικών η Επιτροπή μας θα αποφασίσει. Η τελευταία απόφαση ήταν ότι οι συστάσεις θα έπρεπε να, προκύψει μόνο, να προκύψουν μόνο από τα μέλη της αποστολής. Από ό,τι καταλαβαίνω, η γραμματεία της Επιτροπής μας ε, θα ήθελε όλα τα μέλη της Επιτροπής να μπορούσαν να υποβάλουν συστάσεις. Αν ε, συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ας πούμε ότι 26 Ιουνίου θα ήταν η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για να ψηφίσουμε στην επόμενη, ε, στη συνεδρίαση που θα ακολουθήσει. Συναντήσαμε πολλούς ε, οργανισμούς στο Βερολίνο. Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή με ε, άτομα τα οποία επλήγησαν από την ε, κατάσταση αυτή. Ε, ελπίζουμε όμως ότι ως ευρωβουλευτές είμαστε σε θέση να συζητήσουμε αυτό το θέμα με τις γερμανικές ε, αρχές. Βέβαια με πλήρη σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας δεν θέλουμε να μπούμε στα χωράφια ε, εσωτερικών θεμάτων καμιας χώρας. Ε, να ευχαριστήσω την κυρία Μπομπίνσκα και τους υπόλοιπους συναδέλφους που ήταν εκεί για τις συστάσεις και τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιο το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση και ένα σχόλιο. Καταρχήν, εδώ, μαζί με το σχετικό έγγραφο, έχω και κάποιες τροπολογίες, ε, κάποιες τροποποίησεις προτείνονται από τον κύριο Μπουλάν, που όμως δεν είναι εδώ. Πρέπει να αποφασίσουμε όμως ε, Επίσης, ε, έχω και ένα email της κυρίας Μπομπίνσκα με κάποιες προτάσεις ε, και συστάσεις. Έτσι λοιπόν, ε, θα ήθελα να ρωτήσω τη συνάδελφο πώς προτείνεται να προχωρήσουμε με όλα αυτά τα έγγραφα. Γιατί έχουμε δύο έγγραφα τα οποία είναι εντελώς αντίθετα το ένα με το άλλο. Και να κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με το ποιος μπορεί να συμμετέχει και να δεχτεί τις συστάσεις μας. Εμένα με ενδιαφέρει να συμμετάσχω στην αποστολή αυτή, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό το ζήτημα και με απασχολεί ιδιαίτερα. Ασχολούμαι ιδιαίτερα με αναφορές, με τη χρήση της γλώσσες και υπήρχε και μία παρόμοια συζήτηση κατά χώρες όπου μία οικογένεια από τη Λετωνία κατηγορήθηκε επειδή χρησιμοποιούσε ε, τη γλώσσα της, τη δημητρική γλώσσα εντός της οικογένειας και για το λόγο αυτό πήραν τα παιδιά από την οικογένεια. Δηλαδή τους είπαν δεν μιλάτε Ολλανδικά στην οικογένεια και μιλάτε τη μητρική σας. Αυτό όμως είναι εντελώς απαράδεκτο. Εγώ δεν μπορούσα βέβαια να συμμετάσχω τελικά σε αυτήν την επιστολή γιατί είχαμε και μία αποστολή στη Μολδαβία αν θυμάστε ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν, εσεί ε, πήγατε στο Βερολίνο, εγώ ήμουν στο Κισινάου, αλλά αυτό δεν με εμπόδισε από το να συμμετέχω στη λήψη αποφάσεων. Γιατί όταν ε, ήρθαν οι αναφέροντες στο Κοινοβούλιο και παρουσίασαν ε, αυτέ τι αναφορέ κατά της Jugendamt, εγώ συμμετείχα. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να μην συμμετέχει ποιος δεν μπόρεσε να είναι και στις αντιπροσωπείες. Ευχαριστώ κύριο Γιάρ. Ευχαριστώ για όσους συμμετείχαν σε αυτήν την αποστολή και την εισηγήτρια. Μπορώ να πω ότι μάθαμε κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού Έχω κάνει δύο εκθέσεις για τέτοιου είδους ε, αποστολές και για τη Ρουμανία και για το Βερολίνο και προκύπτει ότι πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο αλλά και περισσότερη ταχύτητα. Πρέπει να καθορίσουμε βέβαια και τη διαδικασία και νομίζω ότι το ελάχιστο στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι συμμετέχονται σε τέτοιου είδους ταξίδια μαζί με την Γραμματεία να κάνουν μια έκθεση βεβαίως και η Επιτροπή, όλα τα μέλη δηλαδή της Επιτροπής, να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τροπολογίες και να γίνεται ψηφοφορία στην Επιτροπή. Γιατί το θέμα είναι ποιος έχει την τελική πολιτική ευθύνη, την τελική πολιτική ευθύνη την έχει η Επιτροπή. Αλλά θέλω να καθησυχάσω τους συναδέλφους. Αυτό βεβαίως σημαίνει απλώς ότι τα μέλη της Επιτροπής μας να κάνουν συστάσεις. Αυτή είναι η διαδικασία. Πρέπει να υπάρχει προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και μετά πρέπει να γίνεται ψηφοφορία. Νομίζω πως θα ήταν δίκαιο αυτό για όλα τα μέλη. Εφόσον ε, γίνονται, γίνονται τέτοιου τύπου αποστολές οι συνάδελφοι που πηγαίνουν τα μάτια και τα αυτιά της Επιτροπής για να συλλέξουν λεπτομεριακή ενημέρωση ούτως ώστε η Επιτροπή μας να είναι σε θέση να εξάγει συμπεράσματα και να ε, μπορεί να κάνει και τις αναγκαίες συστάσεις. Μετά να υποβάλλονται τροπολογίες, μετά να γίνει ψηφοφορία και αυτό το κείμενο θα ε, εκπροσωπεί και θα είναι έτοιμο με την ευρεία έννοια της λέξης για όλους μας. Βέρτμαν. Για δύο σημεία να μιλήσω. Το αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης είναι πολύ σαφές. Πρώτα απ' όλα περιγράφει την κατάσταση. Δεν θα πρέπει να κάνει αξιολογικές κρίσεις ούτε να καταδικάσει. Θα πρέπει να περιγράφει την κατάσταση. Οπότε, επειδή εγώ θα ήθελα, όπως και πολλοί άλλοι πιστεύω, αντικειμενικότητα, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Σε ποιες ε, περιπτώσεις απαγορεύεται εντό εισαγωγικών η χρήση της μητρικής γλώσσας. Από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι είδα στην Επιτροπή μας, αυτό γίνεται μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει όντως κίνδυνος απαγωγής. Και γίνεται για λόγους προστασίας των μικρών, ε, πολλές φορές ε, μικρών παιδιών, πολύ μικρών παιδιών, σταματούν λοιπόν ε, τη συζήτηση και λένε ότι εγώ που είμαι εκεί για να παρακολουθήσω την υπόθεση από πλευρά των αρχών πρέπει να μπορώ να καταλάβω τη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των παιδιών. Και αυτό το λέω και ως μητέρα και πολλοί άλλοι το λένε. Φυσικά οι γονείς πρέπει να μπορούν να μιλάνε στα παιδιά τους, αλλά η προστασία των παιδιών είναι το υπέρτατο καθήκον. Δεν μπορούμε εμείς ως πολιτικοί να αποφασίζουμε για την ε, τύχη και την ευημερία παιδιών που δεν γνωρίζουμε, που δεν γνωρίζουμε τα προηγούμενα και ποια γλώσσα μιλάνε ακριβώς στο σπίτι οι γονείς με τα παιδιά. Αυτό δεν το ξέρουμε. Μπορεί να μιλάνε την ε, μητρική γλώσσα, αλλά σε αυτές τις επισκέψεις όπου έρχονται εκπρόσωποι της αρχής για την νεότητα πρέπει να μπορεί να γίνεται κατανοητή συζήτηση. Γιατί υπάρχει αυτή η επίσκεψη όμως. Πρέπει να είμαστε απόλυτα αντικειμενικοί. Άτομα που δεν ήταν παρόντα. Οι συνάδελφοι που δεν ήταν παρόντες βεβαίως πρέπει να μπορούν να εκφραστούν, βεβαίως πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν θέση, αλλά μόνο με σαφή διαφοροποίηση για θέματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκε η αναφορά και το περιεχόμενό της. Σωστά υπόθηκε. Όταν πηγαίνουμε σε μια τέτοια αποστολή είμαστε τα μάτια και τα αυτιά της Επιτροπής μας. Οπότε, επειδή αυτές οι υποθέσεις είναι πολύ λεπτές, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την απόλυτη αποτελεσματικότητα και δίκαιη αντικειμενική συμπεριφορά. Σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη τις σκέψεις μου αυτές ε, περαιτέρω. Ευχαριστώ την κυρία Φέρτμαν και τον κύριο Μπουστινάρου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι είναι κάπως ντροπιαστικό να βλέπουμε ότι δεν έχουν ψηφιστεί ακόμη δύο εκθέσεις. Και ειλικρινά ήθελα να σας πω ότι περισσότερο είναι θέμα του ΕΛΚ παρά θέμα που εμπλέκει την Επιτροπή ως Επιτροπή. Και η δική μου πρόταση είναι η έκθεση να καταρτιστεί σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θα αποφασιστεί, θα το συζητήσουμε μάλλον αυτό στη συνέδριση των συντονιστών σήμερα και κατόπιν ε, κανένα από τα μέλη της διερευνηστικής αποστολής ή της Επιτροπής θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να ε, παραβιάσει τις χρονικές προθεσμίες. Όταν θα έχουμε θέσει εμείς ε, προθεσμίες για την κατάθεση τροπολογιών, κατόπιν θα πρέπει και να τις σεβαστούμε. Όταν ε, έχει εξαντληθεί ο χρόνος, είτε θα γίνει αποδεκτή τροπολογία, είτε θα απορριφθεί. Και αν απορριφθεί, θα πρέπει να τη βάλουμε στο παράρτημα, όπως κάναμε σε μία από τις δύο εκθέσεις που ανέφερα προηγουμένως. Αλλά Διαφορετικά μπαίνουμε σε διέξοδο. Γιατί κάποιοι από εμά μπορεί να θέλουν τόσο πολύ να επιβάλλουν τη δική τους τροπολογία. Όμως αυτός δεν είναι ο βελτιστός τρόπος ε, για να είμαστε αξιόπιστοι. Αυτή είναι η έκκληση που απευθύνω και θα σταματήσω εδώ. έχοντα κατά νου ότι τελικά οι διερευνητικές αποστολέ θα πρέπει να καταλήγουν σε εκθέσει που να εκφράζουν την πραγματικότητα που είδαμε επί τόπου. Λιγότερο πάθος, λιγότερη πολιτική αντιπαράθεση και αν όχι συνένεση θα έχουμε περισσότερους συμβιβασμούς όπου θα μπορούν να γεφυρώνονται όλες οι θέσεις για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Επιτροπή Αναφορών. Ευχαριστώ. Δεν άκουσα τι είπε η κυρία Γιώτοβα, γιατί καθυστέρησα να έρθω. Όμως φανταζόμαι ότι είπε εδώ σας συμφωνήσαμε. Εγώ νομίζω ότι καθυστέρησε πολύ η έκθεση αυτή για θέματα που συζητούμε και ε, ε, προκειμένου να σεβαστούμε και τους αναφέροντες ε, νομίζω ότι πρέπει επιγόντως να ψηφίσουμε πριν το καλοκαίρι Συμφωνήσαμε ότι τον Ιούλιο θα έχουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Εγώ το προσυπογράφω αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα του ΕΛΚ. Νομίζω ότι κυρίως ε, προσκρούμε σε μία μη ρύθμιση σε ό,τι αφορά τις διερευνητικές αποστολές. Και για το θέμα αυτό υποβάλλω μία πρόταση που ίσως ε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα προβληματισμό για να ρυθμίσουμε τις μελλοντικέ διερευνητικές αποστολές και κάτι τέτοιο να μας επιτρέψει να αποσαφηνίσουμε και τη μέθοδο και τις προθεσμίες ε, της ε, εκπόνησης της έκθεσης. Επίσης λυπάμαι που αλλάξει σκεπτικό γιατί στην αντιπροσωπεία που πήγε στο Βερολίνο είχαμε ψηφίσει κάτι που έπρεπε να γίνει σεβαστό. Έπρεπε να συνεχίσουμε σε εκείνη την οδό. Είχαμε ένα κείμενο επί το οποίο δεν αντιτίθεμε καθόλου, γιατί ούτω ή άλλω ε, εκεί συμπεριλαμβάνονται οι προτάσει που είχαμε υποβάλει, αλλά επί τη μεθόδου ε, νομίζω ότι πρέπει πολύ γρήγορα να προσδιορίσουμε ποια είναι η μέθοδος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για όλες τις ε, διερευνητικές αποστολές Τι κατά θα επιτρέψει σε όλα τα μέλη της Επιτροπής να τοποθετηθούν επί των προτάσεων. Εγώ θα πρότεινα να έχουμε δύο μέρη. Καταρχήν ε, κάτι ε, που θα είναι πραγματιστικό, δηλαδή να έχουμε την σύνοψη της αποστολής ε, όπως υλοποιήθηκε και θα έχουμε και ένα δεύτερο μέρος και εκεί θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι είναι μέλη εξοφίσιο της αποστολής να μην έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων, δεν μπορούν να είναι συντονιστέ, παραδείγματο χάρη. Έτσι λοιπόν, ε, νομίζω ότι ε, με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να σεβαστούμε τι προθεσμίε για τι υπόλοιπε διερευνητικέ αποστολέ. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο έχει μεγάλες διαστάσεις ε, και έχει δραματικές διαστάσεις, αφορά δεκάδες οικογένειες, αν δεν είναι περισσότερες και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό τον Ιούλιο. Όλοι έχουμε αυτή την επιθυμία. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Μπολάνο. Δεν ε, ζητά κάποιο άλλος ε, το λόγο. Κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ. Προτείνω, ακούγοντας ε, τους προηγούμενους, προτείνω σήμερα λοιπόν στις συνεδρίες των συντονιστών να καθορίσουμε προθεσμία για υποβολή τροπολογιών στο αρχικό κείμενο που ήδη παρουσιάσαμε και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μπουρλάν να μου πει αν θα ήθελε να διατυπώσει τις τροπολογίες με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ανταποκρίνονται ε, στον κανονισμό τα άρθρα για τροπολογίες πώς υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρίτον, Καλωσορίζω την ε, επιθυμία όλων των μελών της Επιτροπής μας να υποβάλουν τροπολογίες. Οπότε πρέπει να καθορίσουμε προθεσμία για την ε, υποβολή τους, αλλά και για τη συζήτησή τους. Και εργάστηκα για την έκθεση αυτή δύο μήνες και διάφοροι συνάδελφοι ε, μου έδωσαν την εντύπωση ότι θα ήθελαν να, να η συζήτηση, να καθυστερήσει η διαδικασία και επέμειναν συνεχώς ότι είναι εσωτερικό γερμανικό θέμα και ότι δεν εμπίπτει ε, ε εντός των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες ε, στρέφονται προς την Επιτροπή μας για δικά τους θέματα, της χώρας τους και πρέπει να ε, δώσουμε συνέχεια ε, στις αναφορές τους, στο βαθμό βεβαίως που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας. Όσον αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Μπουρλάν, πρέπει να τονίσω ότι ένας Γερμανός εκπρόσωπος ε, άσκησε πιέσεις για να τροποποιήσω το κείμενο. Αυτό θεωρώ πως είναι εντελώς απαράδεκτο. Θα πρέπει να αντιδράσουμε με κατηγορηματικό τρόπο. γίνει ένα τμήμα αυτής της εργασίας ε, και τον Ιούλιο. Ε, η γραμματεία μας έχει προτείνει και την 26η Ιουνίου ως προθεσμία για να έχουμε και τις μεταφράσεις και κατόπιν προσυπογράφω όσο είπαν κάποιοι συνάδελφοι σε σχέση με το δικαίωμα τα μέλη αυτής της Επιτροπής να παρουσιάζουν τροπολογίες και κατόπιν ε, η Ολομέλη της Επιτροπής θα αποφασίσει αν είναι κατάλληλες αυτές τις τροπολογίες ε, και αν θέλει να τις δεκτεί να τις απορρίψει. Τώρα, σε σχέση με το χρόνο και με το τρόπο κατάρτισης των εκθέσεων για τις διερευνητικές αποστολές, εγώ νομίζω ότι θα κριθούν βάσει ε, της ε, λογικής του καθένα. Θα το δούμε αυτό το σημείο και με τους συντονιστές. Ε, εμείς θεωρούμε ότι αν δεν σεβόμαστε τους κανόνες, θίγει την αξιοπρέπεια του Κοινοβουλίου. Υπάρχει και ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το ΕΛΚ και λυπάμαι για την ειδική μου ομάδα. Ελπίζω να μην ισχύει ε, το θέμα έτσι όπως το παρουσίασε ο κύριος Μπουλάν και στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουλίου ε, ελπίζω όχι μόνο η έκθεση για την αποστολή στο Βερολίνο αλλά και η έκθεση για την αποστολή στην Ρουμανία να μπορούν να οριστικοποιηθούν γιατί όπως είπε και κάποιος σε πρόσφατη παρέμβαση, σε λίγο καιρό θα έχει περάσει ένας χρόνος ε, από τη στιγμή υλοποίηση των δύο αυτών επισκέψεων. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι επισκέψεις θα έπρεπε να χρησιμεύουν για να επιταχύνουν μέσω της συλλογή ε, περαιτέρω πληροφοριών, ε, το πώς θα προχωρούν τα πράγματα στην δική μα επιτροπή. Όμως, μου φαίνεται ότι εμείς τελικά κάνουμε το αντίθετο. Όπω και να έχει, σας ευχαριστώ και ολοκληρώνονται εδώ οι εργασίες ε, του σημερινού πρωινού για να δώσουμε τώρα και τη δυνατότητα στους συναδέλφους και στο κοινό να εγκαταλείψει την αίθουσα και να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών.